Ja, Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ο κύριος Μπουτικόφερ ε, φαίνεται και καλοξυγισμένος, καλοκουρεμένος, κερδίζει το διαγωνισμό. Ναι, τα κατάφερα, είναι πριν από τα Χριστούγεννα, ωραία. Καλώς ήρθατε όλοι. Ε, έχουμε κατόπιν αιτήματο τη Γραμματεία, ένα θέμα το οποίο πρέπει να συζητήσουμε μετά και από τη συζήτηση με τους συντονιστές γιατί πρέπει να ξεκαθαρίσουμε αυτό το θέμα να το κάνουμε όπως συνήθω, όχι μόνο με γραπτή ανακοίνωση Χτες κάναμε τη συνάντηση των συντονιστών που ήταν σύντομη Μιλήσαμε για τον τρόπο εργασιών μας για το συνολικό πακέτο για τον ορίζοντα 2020. Συμφωνήσαμε ότι θα πρέπει να συζητηθούν στην ομάδα εργασίας όλα αυτά που έχουν σχέση με τους εισηγητές και σκιώδεις εισηγητές και θα πρέπει να ληφθεί απόφαση στην Ολομέλεια το φθινόπωρο του 2012. Ε, θέλουμε να συζητήσουμε τμήματα αυτού του πακέτου το συντομότερο δυνατόν. Υπήρχαν ε, πολλές ε, προτάσεις και δεν καταλήξαμε σε κάποια συγκεκριμένη απόφαση του επόμενου σημείου και μετά για το θέμα της κατανομής των εκθέσεων πάλι δεν προχώρησε πάρα πολύ το θέμα διότι η διαδικασία την οποία έχουμε όταν ανακοινώνονται εκθέσεις στην Ολομέλεια είναι μια διαδικασία την οποία δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε ε, ε, τίποτα γιατί είναι ο ασφαλέστερος τρόπος στον οποίο και παραμένουμε. Δώσαμε, ε, αναθέσαμε τις εκθέσεις για τον ορίζοντα 2020. Στη βασική έκθεση την ανέλαβαν οι σοσιαλιστές, κανόνες συμμετοχή στο ΕΛΚ. Μετά είχαμε στρατηγική καινοτομία πήρε η Γκουε ε, και μετά τροποποίηση του κανονισμού που πήραν οι πράσινοι ε, υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Δορυφόρου πήρε το ΕΛΚ πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων πήραν οι φιλελεύθεροι και μια τροποποίηση της οδηγίας ε, ε, για την, χρησιμοποίηση των ε, πληροφοριών του δημοσίου τομέα οι σοσιαλιστές και κάποιες γνωμοδοτήσεις αγορά και χρηματοοικονομικά εργαλεία το δεύτερο τμήμα πήρε το, πήραν οι φιλελεύθεροι προγράμματα περιβάλλοντος και live το ΕΛΚ πρόγραμμα για τη δημιουργική Ευρώπη οι σοσιαλιστές νοτόμα χρηματοπιστωτικά εργαλεία στο πλαίσιο του πολιετούς δημοσιονομικού προγράμματος, το ΕΛΚ. Οπότε τώρα σας ενημέρωσα για όλα όσα έγιναν χτες και τουλάχιστον εσείς που είστε παρόντες τώρα γνωρίζετε. Το πρώτο σημείο για σήμερα το πρωί τώρα είναι το σημείο 6, Ευρωπαϊκή Τυποποίηση. Ο συνάδελφος Γκίρεκ είναι εισηγητής και του δίνω κατευθείαν το λόγο. Κύριε Γκίρεκ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κανονισμός ε, του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου που συζητούμε σήμερα έχει ως στόχο να επηρεάσει θετικά τις διαδικασίες ε, της ε, αγορά σε ό,τι αφορά την καινοτομία, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα. Στόχος λοιπόν είναι η διαδικασία τυποποίησης ε, να είναι πιο σύντομη και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να εκπροσωπούνται κατάλληλα ως μελλοντικοί εμπλεκόμενοι φορείς σε αυτή τη διαδικασία τυποποίησης. Επίσης θα πρέπει να διαδίδονται τα πρότυπα στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και των τεχνολογιών. Και μέσω αυτής της διάδοσης στόχος είναι και η βελτίωση της διαλειτουργικότητας. από ό,τι φαντάζομαι γνωρίζετε, υπάρχουν πολλά προβλήματα με τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων πληροφορικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα άλλο θέμα είναι κάτι που συχνά παραβλέπετε και συγκεκριμένα είναι τεχνολογίες, οι βιοτεχνολογίες, η πυρηνική τεχνολογία και τα σχετικά. Οι μείζονες αλλαγές ε, στην πρόταση κανονισμού έχουν να κάνουν ε, με τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της μόνιμης επιτροπής για τα πρότυπα, το Standing Committee. Περιλαμβάνει επίσης την τυποποίηση στις υπηρεσίες καθώς και μία ξεχωριστή μεταχείριση για τη δέσμη των τεχνολογιών των πληροφοριών. Έγινε επίσης και αλλαγή ε, στη χρηματοδότηση, στη διαδικασία χρηματοδότησης. Ως ε, εισηγητής είμαι υπέρ της πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου και, της, ε, και του Κοινοβουλίου, γιατί νομίζω ότι θα παγιώσει την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της τυποποίησης, ενώ εισάγει και νέα στοιχεία τα οποία θα μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις. Άρα με τον τρόπο αυτό μπορούμε να εξυγχρονίσουμε την ε, ενιαία αγορά, βελτιώνοντας και το ευρωπαϊκό σύστημα τυποποίησης. Σύστημα κοινοποίησης προτύπων για υπηρεσίες και συγκεκριμένα ηλεκτρονικές. Επίσης θα πρέπει να μιλήσουμε για τη χρηματοδότηση των προτύπων. Αυτό το προανέφερα Υπάρχει τώρα μια καλύτερη νομική βάση για τη χρηματοδότηση της Κομισιόν και για την απλούστευση επίσης της διαδικασίας τυποποίησης. Βέβαια, υπάρχουν κάποιες ανησυχίες σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα ορισμένων διατάξεων του κανονισμού. Συγκεκριμένα, ε, συμπράξεις σε ε, ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Θα πρέπει ο κανονισμός να συνταχθεί κατά τρόπο ώστε να αποτελεί συνάμα και ένα εφαρμοστικό εργαλείο που θα αποσκοπεί στην πρόθεση της ε, νέας αγοράς και στην εφαρμογή ευρωπαϊκών προτύπων για να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα και η συμμετοχή των ε, εμπλεκομένων μερών, αλλά και η βιώσιμη ανάπτυξη. Άρα το σύστημα τυποποίησης πρέπει να βελτιωθεί με την εισαγωγή αυτών των νέων στοιχείων. Τα στοιχεία αυτά μάλιστα θα συνιστούν προστιθέμενη αξία Έρχομαι τώρα σε κάποιες ειδικότερε παρατηρήσεις. Δεν αναφέρονται ισχύωτες κανόνες της ευρωπαϊκής τυποποίηση. Παραδείγματο χάρη, εθνική εκπροσώπηση ως αρχή δεν αναφέρεται. Ούτε η αρχή του status quo, stand still, αναφέρεται μια αρχή ουσιαστική σημασία για την εναρμόνιση των προτύπων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει εναρμόνιση. Πολλές διατάξεις επίσης είναι γενικόλογες. Σε ό,τι αφορά παραδείγματο χάρη την εκχώρηση εξουσιών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιτρέπει αυτό πολύ ευρία ερμηνεία των διατάξεων και συγκεκριμένα σε τομείς που προτείνονται αλλαγές για τη λειτουργία του ισχύοντος συστήματος. Προτείνονται επίσης αυτό το σχέδιο μια σειρά από τεχνικές προδιαγραφές Μια από τις βάσεις της δημοκρατικής διαδικασίας τυποποίησης είναι η κοινωνική συνένεση. Η ακαιρεότητα του ευρωπαϊκού συστήματος τυποποίησης είναι η δύναμή του καθότι διασφαλίζει τη συνοχή μιας δέσμης προτύπων. Η συμμετοχή φόρουμ και κοινοπραξιών στο σύστημα δεν πρέπει να οδηγήσει στον καθορισμό αντιφατικών προτύπων και ανταγωνιστικών μεταξύ τους προδιαγραφών, ούτε και να παρεμποδίζει τη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και, τα έξοδα συμμετοχή σε φόρουμ είναι υψηλά, τα κριτήρια τύληψη των αποφάσεων δεν είναι πάντοτε δημοκρατικά. Επίση, ορισμένα φόρουμ και κοινοπραξίε ενδέχεται να κυριαρχούν παράγοντε εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Ω εκ τούτου, καλό θα ήταν η εκπόνηση προτύπων να περιορίζεται στους αναγνωρισμένους σήμερα Ευρωπαϊκού Οργανισμού τυποποίηση ενώ θα πρέπει να αξιοποιηθούν οι πολυάριθμες δυνατότητες που προσφέρονται από τους οργανισμούς αυτούς προς την εκφώνηση εγγράφων βάση επίγουσας βασινό, βασιζόμενης σε συνένεση διαδικασία στην οποία θα λαμβάνουν μέρος ενδιαφερόμενοι παράγοντες από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει να εφαρμόζονται σε αυστηρά προσδιορισμένες περιπτώσεις. Οι απαιτήσει δεν πρέπει να είναι πάντα ίδια. Συνένεση, δημοσιότητα, θελοντική συμμετοχή, διαφάνεια και ούτω καθεξής. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών, θα πρέπει να εγγυηθούμε και εδώ τη διελειτουργικότητα. Είναι αξιέπαινος ο στόχος, όπως είπα και στην αρχή. Υπάρχουν όμως δυσκολίες. Πώς θα πετύχουμε τους στόχους αυτούς. Το έγγραφο προτείνει έναν μόνο τρόπο. Και ίσως να μην είναι το βασικό μονοπάτι, το κυριότερο που θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε. Είναι πάντως ένας δρόμος ο οποίος θα μας επιτρέψει να επιταχύνουμε τις διαδικασίες αυτές. Επίσης θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε καλύτερα τα διάφορα φόρουμ κατά την εκπόνηση ή πριν την εκπόνηση δια, ε, κανονισμών για τις τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών. Υπολείπεται κατά κάποιο τρόπο θα έλεγα σε αυτό τον τομέα Ευρωπαϊκή Ένωση. σε σχέση με τους ανταγωνιστές της. Ε, αυτά είχα να πω, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον εισηγητή. Θα δώσουμε τον λόγο στην Επιτροπή τώρα πρώτα για να μας παρουσιάσει την έκθεση. Κυρία Μπρίκμαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δίνετε στην Κομισιόν την ε, δυνατότητα να παρουσιάσει στα μέλη της Επιτροπής σας τα κυρία στοιχεία της πρότασής μας, επικεντρωνόμενη στα θέματα των αρμοδιοτήτων μας. Και θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Γκίρεκ για την υποστήριξή του για την πρότασή μας. Σημειώσαμε τα διάφορα στοιχεία της, ε, που εξέφρασε στην εκθεσή του. Εδώ θα προσπαθήσω στην παρουσίασή μου να αναφερθώ στα περισσότερα στοιχεία και να απαντήσω στα περισσότερα στοιχεία που ανέφερε ο κ. Γκίρεκ. Και θα σας εξηγήσω γιατί έχουμε κάνει την πρόταση που έχετε σε αυτή τη στιγμή. Καταρχήν, να σας εξηγήσω ότι πρόκειται για δέσμη μέτρων, δηλαδή δεν μιλάμε μόνο για κανονισμό, αλλά και για ανακοίνωση. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί στον τομέα της τυποποίησης δεν χρειαζόμαστε νομοθετήματα για όλα τα στοιχεία της στρατηγικής. Και γι' αυτό Παρουσιάσαμε το πακέτο με μια ανακοίνωση όπου αναφέρεται το στρατηγικό όραμα για την τυποποίηση μέχρι το 2020 και ένα νομοθέτημα το οποίο συνοδεύει την ανακοίνωση. Αυτό είναι σημαντικό γιατί ορισμένα στοιχεία από τα οποία ανέφερε ο κύριος Γκίρεκ που δεν βρίσκει στον κανονισμό όντως δεν είναι στον κανονισμό, αλλά εξηγούνται στην ανακοίνωση. Θα ήθελα λοιπόν να σας εξηγήσω ότι έχουμε τώρα τον κανονισμό και το μεγαλύτερο όφελος είναι ότι εφαρμόζεται απευθείας στα κράτη-μέλη, δεν χρειάζεται μεταφορά στο εθνικό δίκαιο. Και... Επίσης, καλύπτει και τις απαιτήσει της Κομισιόν αλλά και τους φορείς της Ευρωπαϊκής Τυποποίησης. Στον ενό κανονισμό θα βρείτε όλα τα στοιχεία που σε αυτή τη στιγμή έχουμε σε διάφορα νομοθετήματα. Έτσι λοιπόν είναι πιο φιλικό προς το χρήστη και σε ένα και μόνο κείμενο μπορείτε να βρείτε όλα τα στοιχεία που χρειάζονται για την εφαρμογή του κανονισμού. Στις διαφάνειες, λοιπόν, βλέπετε τα διάφορα νομοθετήματα που θα αντικατασταθούν, θα αντικατασταθούν εν μέρη. Θέλω κάτι που θέλω να αναφέρω συγκεκριμένα για την οδηγία 9834. Επιμένουμε ότι εδώ μιλάμε για την τυποποίηση και όχι για τεχνικό κανονισμό. Το τμήμα που έχει να κάνει με τον τεχνικό κανονισμό στην 9834 δεν φύγεται καθόλου από τη δική μας πρόταση. Δεν μιλούμε λοιπόν εδώ για τεχνικό κανονισμό, μιλούμε μόνο για πρότυπα. Και όπως ξέρετε είναι το 834 έχει να κάνει και με τα δύο αυτά. Αυτό είναι σημαντικό γιατί δεν μιλάμε για πρότυπα, το όραμά μας είναι ότι μιλάμε για ιδιωτικά μέσα για τον τομέα και είναι εκούσιο χαρακτήρα, δεν είναι υποχρεωτικά όπως ο κανονισμός. Να δούμε την επόμενη διαφάνεια. Σε πολλές περιπτώσεις είπαμε ότι αυτό που προτείνουμε είναι μια εξέλιξη και όχι επανάσταση και θέλουμε να σας πούμε περί τίνος πρόκειται. Δεν αλλάζει το σύστημα, δεν αλλάζει η φύση των προτύπων, ε, Έκουσε χαρακτήρα, προσέγγιση, δύναμη των αναγκών της αγοράς. Ε, επιμένουμε πάντα στην υπεροχή των διεθνών προτύπων, δεν υπάρχει αλλαγή για το ρόλο των ευρωπαϊκών φορέων τυποποίησης. Δεν αλλάζουμε τίποτα για το ρόλο των φορέων αυτών των οργανισμών τυποποίησης. Θα ξέρετε ότι η Κομισιόν έχει δώσει ένα μοναδικό καθεστώς ε, σε αυτούς τους οργανισμούς, δηλαδή τους δίνει μια προνομιούχο θέση για την εκμόνηση των ευρωπαϊκών προτύπων. Έχουμε αυτή την ε, συμφωνία, εταιρική συμφωνία πλαίσιο Συμφωνία Εταιρική Σχέση και χρηματοδοτούμε το κόστο μέχρι 50%. Πρόκειται για ιδιωτικέ οργανώσει δηλαδή, αλλά έχουμε ειδική σχέση με αυτέ. Και γι' αυτό έχουμε εισαγάγει στοιχεία σε σχέση με το είναι αναφορά σε αυτούς τους οργανισμούς ε, στον ίδιο τον κοινωνισμό τυποποίησης. Ε, επίσης ε, δεν αλλάζει η αρχή της εθνικής εκπροσώπησης και δεν αλλάζουμε τίποτα σε σχέση με την ε, εντολή των ΕΣΟ, των οργανισμών τυποποίησης. Αυτά τα διατηρούμε άθικτα στον κανονισμό. Δεν θα βρείτε αυτό το στοιχείο, θα το βρείτε στην ανακοίνωση, γιατί ένα νομοθέτημα πρέπει να σέβεται αυστηρά κριτήρια και δεν ε, είναι στοιχεία που μπορείτε να βρείτε στον κανονισμό αυτά, γι' αυτό τα αναφέρουμε στην ανακοίνωση και εκεί εξηγούμε πλήρως όλο το σύστημα που αποτελεί τη βάση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Τυποποίησης στην Ευρώπη, το οποίο δεν τροποποιείται όπως σας είπα. Ο σας αναφέρω μια σειρά καινοτομιών. Θα ήθελα να δω και εγώ, να δούμε μαζί τη καινοτομία του κανονισμό. Καταρχήν, η Κομισιόν, μετά από διαβούλευση με τα διαφορεμένα μέρη, θα εκπονήσει ένα ετήσιο πρόγραμμα εργασία. Αυτό θα βασίζεται σε ανοιχτή διαβούλευση και σε έναν με όλες τα ενδιαφερόμενα μέρη. Προ στιγμή δεν έχουμε αυτό το ετήσιο πρόγραμμα. Προετοιμάζουμε ένα, το οποίο θα υιοθετηθεί από την Κομισιόν τις επόμενε εβδομάδες και αυτό θα σας δείξει πως ε, τα ευρωπαϊκά πρότυπα υποστηρίζουν όχι μόνο την ευρωπαϊκή νομοθεσία αλλά και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν ε, για να υποστηρίξουν τις κυρίες θεματικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως ε, η σύμπραξη για την κεντομία, το ψηφιακό θεματολόγιο, το Resource Europe έτσι λοιπόν βλέπετε ποιε εντολέ σκοπεύει να δώσει η Κομισιόν για του χρόνου. Πρόκειται για μια πρώτη δοκιμή. Δηλαδή να παρουσιάσουμε στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο τις προτεραιότητες για το πρόγραμμα εργασίας για τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Αυτό το πρόγραμμα εργασίας αναφέρεται στον κανονισμό γιατί είναι πολύ σημαντικό νέο στοιχείο και θα πάρει τη μορφή ανακοίνωση προς το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Ο εισηγητής ε, ανέφερε και την επέκταση της υπηρεσίας, αλλά εδώ θέλουμε να επιμείνουμε στο ότι όπως και για τα αγαθά, θα προτείνουμε επέκταση στον τομέα των υπηρεσιών μόνο αν υπάρχει δημόσιο ενδιαφέρον και έτοιμο από την αγορά. Έτσι λοιπόν η φύση των προτύπων δεν διαφέρει, χρησιμοποιούμε την ίδια αρχή. Θέλουμε να έχουμε και ένα πιο συμπεριληπτικό σύστημα για την ε, προωθημένη συμμετοχή των stakeholders. Ε, ανέφερε ο εισηγητής νέες αρμοδιότητες της Κομισιόν, περιέχονται από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Και έχουμε την επιτροπολογία που καθορίζεται δυνάμει της συνθήκης της Λισαβόνας. Αυτό αναφέρεται στην πρότασή μας, ε, διάταξη για τις κατεξουσίες της πράξης και επίση θέλουμε να προβλέψουμε και τη δυνατότητα χρησιμοποίησης ε, των υφιστάμενων προδιαγραφών ε, τεχνολογιών επικοινωνιών και πληροφοριών ε, από τα διάφορα φόρα και τι κοινοπραξίε, τι πολιτικέ και στις προμήθειε. Έτσι λοιπόν, σε αντίθεση με τους οργανισμούς τυποποίησης, δεν θα δώσουμε εντολή στη φόρα και στις κοινοπραξίες να εκμονήσουν πρότυπα στον τομέα των πληροφοριών, πληροφοριών και επικοινωνιών. Δεν έχουμε καμία τέτοια πρόθεση. Ο κανονισμός εξηγεί πώς θα χρησιμοποιήσουμε συγκεκριμένες υφιστάμενες προδιαγραφές ICT, δυνάμεις συγκεκριμένων κριτηρίων που πρέπει να σεβαστούμε. Αυτό το στοιχείο λοιπόν είναι σημαντικό γιατί ενίοτε μπορεί να υπάρχει σύγχυση μεταξύ του ότι δίνουμε εντολή στους οργανισμούς τυποποίησης να εκπονήσουν πρότυπα στον τομέα της τυποποίησης και συγκεκριμένα τομέα των ε, ICT, τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών, θα χρησιμοποιήσουμε τα φυστάμενα, δεν θα δώσουμε εντολή. Έτσι λοιπόν, η εντολή των ε, ΕΣΟΣ, δηλαδή των οργανισμών, Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης, ε, θα παραμείνει ως έχει, δεν θα δώσουμε σε άλλον οργανισμό το ρόλο να εκπονεί ευρωπαϊκά πρότυπα. Αυτό είναι σημαντικό στοιχείο και θέλω να το ξεκαθαρίσω γιατί μπορεί να υπάρχει παρεξήγηση. Τώρα, μικρές και μεσές επιχειρήσεις ε, και ενδιαφερόμενα μέρη. Εδώ θα βάλουμε υπό την ίδια νομική ομπρέλα τους καταναλωτές μικρές και μεσές επιχειρήσεις, ε, τα περιβαλλοντικά και τα κοινωνικά συμφέροντα και επιμένουμε στην εκπροσώπηση, ε, στην ε, εκπόνηση πολιτικής και σε όλα τα κυρία στάδια στη διαδικασία της τυποποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αυτό το βλέπετε στον κανονισμό γιατί και πάλι αναφερόμαστε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε εθνικό επίπεδο επιμένουμε να αρχίσει η ίδια αρχή, αλλά φυσικά αυτό δεν μπορεί να μπει σε ένα κανονισμό, γι' αυτό το έχουμε στην ανακοίνωση. Στην ανακοίνωση μπορείτε να βρείτε Μία από τις ε, δράσεις ε, απαιτείται από τα κράτη-μέλη, δηλαδή να ε, διασφαλίσουν την επαρκή συμμετοχή των stakeholders σε εθνικό επίπεδο. Και επίση προτείνουμε ορισμένα κριτήρια χρηματοδότηση για τι μικρέ και μισέ επιχειρήσει και για τα ενδιαφερόμενα μέρη. Μέχρι τώρα δεν είχαμε εναρμονισμένα κριτήρια. Έτσι λοιπόν όλα αυτά τα ενδιαφερόμενα μέρη θα χρηματοδοτούνται βάσει εναρμονισμένων κριτηρίων. Και επίση ε, θα θέλαμε να έχουμε περισσότερη εκπροσώπηση και ε, αξιμένη ανταπόκριση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης. Αυτό το στοιχείο της πρότασής μας είναι πολύ σημαντικό. Και πάλι για τη θέση των έσω των οργανισμών τυποποίησης. Είναι πολύ σημαντικό να επιμένουμε από αυτό. Σαν σαν έτσι θα συνεχίσουν να έχουν ε, το μονοπόλιο στην εκπόνηση ευρωπαϊκών προτύπων. Αυτό είναι σημαντικό. Το, σύστημα, το ευρωπαϊκό σύστημα προτύπων έχει λειτουργήσει καλά. Και όλοι έχουμε δει ότι τα αποτελέσματα είναι καλά. Θα πρέπει λοιπόν να συνεχίσει να βασίζεται σε αυτή την ειδική σχέση μεταξύ κομισιών και αυτών των ειδικών φορέων, των ιδιωτικών φορέων τι θέλουμε, να έχουμε πιο ξεκάθαρες προθεσμίες για την παραγωγή των αποτελεσμάτων και κάποια χρηματοδότηση βάση των επιδόσεων, αν θέλουμε να εξυγχρονίσουμε, την επιταχύνουμε το σύστημα, χωρίς να θίξουμε τη δομή του συστήματος. Δικαιούμαστε να το ζητήσουμε καλύτερες επιδόσεις. Αυτό θα γίνει μέσω της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης. Θα τροποποιήσουμε την υφιστάμενη και του χρόνου όταν θα ο νέος χρηματοοικονομικός κανονισμός θα εφαρμόσουμε μια νέα τέτοια συμφωνία εταιρικής σχέσης ε, με τους ΕΣΟ, με τους οργανισμούς τυποποίησης, για να λάβουμε υπόψη το περιεχόμενο του νέου χρηματοοικονομικού κανονισμού. Επίσης πρέπει να θέσουμε για κάποιους στόχους έχουμε στόχους αύξησης ε, της αποτελεσματικότητας 50% μέχρι το 2020 και όταν θα έχουμε τον χρηματοοικονομικό κανονισμό, τον δημοσιονομικό κανονισμό και τη νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης θα εισαγάγουμε τα στοιχεία πλούστευσης τα οποία θα συμπεριληφθούν στο νέο χρηματοοικονομικό κανονισμό. Μιλάμε για καταποκοπή ποσά αυτό θα εισαχθεί στην ε, νέα συμφωνία εταιρική σχέση, ε, σύμφωνα με την αθεώρηση και του χρηματοοικονομικού κανονισμού. Ελπίζουμε ότι αυτό μπορεί να γίνει του χρόνου. Επίση, ε, συμπεριλαμβάνουμε και πιο διαφανή υποβολή εκθέσεων με τη συμμετοχή σε εθνικό επίπεδο. Δίνουμε, τους δίνουμε δηλαδή μεγαλύτερο ρόλο, αλλά και τους ζητάμε να επιταχύνουν τη διαδικασία χωρίς ε, φυσικά αυτό να γίνεται σβάρος της ποιότητας των προτύπων. Αλλά φυσικά λαμβάνουμε υπόψη και την ε, αναθεώρηση της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και αν υπάρχει κάποια πλούστευση εκεί θα εκτιμηθεί από τους οργανισμούς ε, τυποποίησης. Υπάρχει ένα θέμα που αφορά το χρονοδιάγραμμα από τη στην έκθεση. Προθεσμία να εκδοθεί εντολή, προθεσμία να απαντήσουμε και να αναθέσουμε μια σύμβαση. Φαίνεται σαν να υπάρχει ανισορροπία. Θέλω να αναφερθώ σε αυτό το θέμα. Μπορείτε να μας μοιράσετε μεγεθυντικούς φακούς για να βλέπουμε. Okay, you don't want that? Too small. I will, I will, I will say it. Okay, I will say δεν βλέπετε καλά, μάλιστα θα τα πω, θα τα πω, μην ανησυχείτε. Στα άρθρο τρία του κανονισμού υπάρχει ένα αίτημα στον κανονισμό, η ΕΣΟ, να απαντήσουν μέσα σε ένα μήνα σε μια προτινόμενη εντολή. Και κατόπιν η Κομισιόν έχει τρεις μήνες για να παράσχει τη σύμβαση. Δηλαδή, Αφενός είναι πιο εύκολο να απαντήσουν οι οργανισμοί τοποποίησης, γιατί θα υπάρχει ανάντηση και διαβούλευση ε, βάσει του ατησίου προγράμματος εργασίας για τη μελλοντική εντολή. Έτσι λοιπόν ε, δεν ε, θα υπάρχει έκπληξη γιατί από την αρχή θα έχουν συμμετάσχει στην εκπόνηση των προτεραιοτήτων. Γι' αυτό λέμε ότι ένας μήνας λογικά αρκεί για να απαντήσουν οι οργανισμοί τυποποίησης γιατί θα πρόκειται για κάτι που θα το γνωρίζουν ε, για μήνες ήδη και θα έχουμε συνεργαστεί για την εκπόνηση των προτεραιοτήτων. Οι τρεις μήνες έρχονται στη συνέχεια και μετά μιλάμε για διάφορα βήματα που σχετίζονται με την αρχή της ε, ορθής δημοσιονομικής διαχείρισης. Παραδείγματο χάρη πρέπει να αξιολογήσουμε τις προτάσεις, αν είναι κατάλληλες, ποιοτικές, να είναι αποτελεσματικές ω προ τον προϋπολογισμό και πρέπει να εκπονήσουμε την πρόταση. Και αυτό σημαίνει ότι έχουμε διάφορα βήματα. Σίγουρα μπορούμε να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τον τρόπο εργασία μα ε, και να εκπονήσουμε τη συμβασή σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά δεν είναι το ίδιο πώς να απαντήσουμε ναι, ναι ή όχι σε μία εντολή. Μπορούμε να επανέλθουμε όμω στο θέμα αυτό. Τώρα το θέμα των προδιαγραφών ICT ε, τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών. Είναι σημαντικό θέμα, όπως είπε και ο συγητής. Υπάρχουν ε, δύο τρόποι εργασία Και πάλι θα βρείτε την εξήγηση στην ανακοίνωση. Ενθαρρύνουμε τη συνεργασία μεταξύ των ΕΣΟ και των φόρουμ και των κοινοπροξιών για την ανάπτυξη των προτύπων αισθητή, αλλά ταυτόχρονα καθώς ε, υπάρχουν ε, πολλές προδιαγραφές που έχουν διευθυνθεί και ε, φυσικά αυτό συμβάλλει στην διαλειτουργικότητα, θέλουμε να παράσχουμε μια δυνατότητα αναγνώρισης των υφιστάμενων προδιαγραφών ICT. Αλλά υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Θα δεχόμασταν ότι μετά από διαβούλευση των ενδιαφερομένων ε, μερών της πλατφόρμας που θα έχει δημιουργηθεί και θα τεθεί σε λειτουργία του χρόνου, το 2012 δηλαδή, θα υπάρχει μια σειρά κριτηρίων. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις εφιστάμενες προδιαγραφές τεχνολογιών, πληροφοριών και επικοινωνιών σε τομείς όπου ήδη έχουμε ευρωπαϊκά πρότυπα. Αλλά θα το πράξουμε μόνο στην περίπτωση που τα ευρωπαϊκά πρότυπα θα είναι πεπελωμένα ή δεν υπάρχουν καθόλου ευρωπαϊκά πρότυπα. Και επίσης ε, θα συμπεριλάβουμε και μια σειρά ποιοτικών κριτηρίων, πολύ αυστηρά κριτήρια. Δηλαδή, καταρχήν, ε, να, γίνεται, να σεβόμαστε τους κανόνες φράντ ε, και τις κατευθυντήριες γραμμές του ανταγωνισμού στις ε, οριζόντιες συμφωνίες συνεργασιών και οι προδιαγραφές ε, θα πρέπει να σέβονται τις αρχές της διαφάνειας, του ανοιχτού χαρακτήρα της συνένωσης κτλ. Και κάτι τελευταίο για τη σημασία αυτού του κανονισμού. Δεν θέλαμε βέβαια να υιοθετηθεί σύντομα και να τεθεί σύντομα σε ισχύ. Πιθανότητα 1η Ιανουαρίου 2013. Όπω είπε και ο εισηγητή, είναι σημαντικό για την ενιαία αγορά, για το ψηφιακό θεματολόγιο και για τι μικρέ και μεσαίε επιχειρήσει. Έχουμε και την ανάγκη να απαντήσουμε στις ε, κοινωνικές προκλήσεις. Και καθώς αυτό το θέμα είναι σημαντικό ήδη το 2013 θα έχουμε μια ανεξάρτητη αναθεώρηση των αλλαγών που έχουμε εισαγάγει. Μια ανεξάρτητη μελέτη των ε, αλλαγών που έχουμε εισαγάγει. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κ. Μπρεζίν έχει ζητήσει το λόγο πρώτος. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με την ε, ε, νομοδότηση του συναδέλφου Γκίρεκ. Έχω συζητήσει και με άλλους συναδέλφους από άλλα κράτη-μέλη και δεν θέλουμε να υπάρξουν σημαντικές αλλαγές. Μόνο κάποια σημεία σε λεπτομέρειες έχω να παρατηρήσουμε. Στην αιτιολόγηση, στην αιτιολόγηση των τροπολογιών, οι 5, οι 6 και οι 8 που αφορούν τα σημεία 19, 20 και 22, εκεί υπάρχει η έννοια της τυποποίησης που τροποποιείται και γίνεται τεχνικές προδιαγραφές. Δεν είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν επαρκείς λόγοι για να γίνει αυτή η τροποποίηση. Τα πρότυπα βασίζονται ε, σε τεχνικούς κανόνες που ισχύουν ε, σε κάθε τομέα και δεν ξεκινούν από τεχνικές προδιαγραφές του κλάδου. Προσπαθήσαμε να ακολουθήσουμε και τις οδηγίες των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης που πολλές φορές ε, διαφέρουν από πρότυπα που προτείνονται από φόρουμ και κοινοπραξίες. Στα υπόλοιπα σημεία της γνωμοδότησης είμαι σύμφωνος. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε ο κύριος Μπιουτικόφερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να προτείνω για την Επιτροπή μας τουλάχιστον να έχουμε ένα πρότυπο για το μέγεθος των χαρακτήρων που θα μας παρουσιάζονται στα slides. Γιατί όταν βλέπουμε τέτοια slides και δεν μπορούμε να διαβάσουμε τίποτα, ε, δεν εξυπηρετεί την ποιότητα της εργασίας μας. Και έχω τρεις παρατηρήσεις τώρα όσον αφορά το θέμα μας. Καταρχήν ευχαριστώ τον εισηγητή για την πολύ προσεκτική δουλειά που έχει κάνει Σας ευχαριστώ ιδίως διότι λάβατε υπόψη σας τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ε, στο πλαίσιο της κοινωνίας των πολιτών, τους societal stakeholders. Η Επιτροπή μας, κατά την ε, τρέχουσα θητεία του Κοινοβουλίου, έχει συζητήσει πολλές φορές το θέμα των οργανισμών τυποποίησης και ε, κατά πόσο προέρχονται από τον τομέα ε, των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων και, της, και των societal stakeholders. Είναι μια συζήτηση που δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Εμείς θα θέλαμε να ενισχύσουμε το ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη διαμόρφωση προτύπων. και στην τροπολογία 18 νομίζω ότι γίνεται μια προσπάθεια για να βελτιωθεί η εκπροσώπηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τώρα όσον αφορά τα πρότυπα από φόρουμ και κοινοπραξίες, είναι ένα από τα βασικά σημεία αυτής της δέσμης μέτρων. Και θα πρέπει να πω ότι η οι ισχυρέ επιφυλάξεις όσον αφορά τα πρότυπα για φόρουμ και κοινοπραξίες που υπάρχουν στη δική σας έκθεση δεν με βρίσκουν απόλυτα ε, σύμφωνο. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να έχουμε πρότυπα και από αυτόν τον τομέα των φόρουμ και κοινοπραξιών δηλαδή. Εσείς προτείνετε κάποιες ε, τροποποίησεις στα άρθρα 9 και 10 και νομίζω ότι ε, με αυτές τις τροπολογίες σας, με αυτές τις τροποποίησεις που προτείνετε εσείς, ε, δεν προωθείτε η συμμετοχή αυτών των φόρμ και κοινοπραξιών και των προτύπων, όπω όπως εγώ θα το επιθυμούσα. Χρειαζόμαστε επίσης το σωστό νομικό πλαίσιο για αυτό τον τομέα παροχής υπηρεσιών και νομίζω ότι εδώ συμφωνούμε όλοι ότι πρέπει να βρούμε τη σωστή οδό και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και σε όλα τα κράτη-μέλη, τουλάχιστον στο δικό μου κράτος μέλος, ε, υπάρχει μεγάλη ανησυχία για τη συμμετοχή ε, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ακριβώς ε, στο συγκεκριμένο τομέα. Εδώ χρειάζεται λοιπόν να ακολουθήσουμε πολύ προσεκτικά βήματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Coffer. Δεν ήσασταν χτες που είχαμε ακόμη πιο μικρά γράμματα στα slides, αλλά έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Θα πρέπει όντως να ζητήσουμε από όλους ε, που κάνουν παρουσιάσεις να μας βάζουν λίγο μεγαλύτερα, μεγαλύτερους χαρακτήρες στα slides. Χτες δεν μπορούσαμε καθόλου να τα διαβάσουμε, ήταν πάρα πολύ μικρά. Συνάδελφος Ούντι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καθώς μιλάμε εδώ για τη σύνταξη και την εκπόνηση των προτύπων, νομίζω ότι θα πρέπει να καταργήσουμε την κοινωνία, γιατί τελικά με όλα αυτά τα αρχικά χανόμαστε και μπερδευόμαστε. Θέλω να υποστηρίξω την ανησυχία του συναδελφού Μπουτικόφερ για τις μικρές και μισές επιχειρήσεις ο συνάδελφος και συνάδελφε κύριε Γκύριακ, δεν καταλαβαίνω τις ε, τροποποιήσεις. Μίλησε ο κ. Μπετικόφερ για την 18 ε, η τροπολογία, αλλά έχουμε και τις τροπολογίες 4 και 19, όπου φαίνεται ότι η συμμετοχή των μικρών και μεσών επιχειρήσεων ουσιαστικά κάπως αποδυναμώνεται. Εγώ νομίζω ότι το αρχικό κείμενο της Κομισιόν ήταν καλύτερο γιατί επιβάλλει την παρουσία των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ε, και ξέρουμε ότι είναι λιγότερο ότι έχουν λιγότερα μέσα από τις μεγάλες επιχειρήσεις για να ακουστεί η φωνή τους. Έτσι λοιπόν πρέπει να τις υποστηρίξουμε και ξέρουμε ότι πρόκειται για ένα τομέα που προοπτικές ανάπτυξης ε, είναι οι πιο ψηλές πιθανότητα. Δεύτερη παρατήρηση, σε σχέση με τις βιομηχανικές ε, πτυχές ε, θεωρώ ότι δεν τονίζεται παρκώς η βιομηχανία Καταλαβαίνω ότι δεν πρόκειται για το μιακό κείμενο, αλλά παρόλα αυτά στο παράρτημα 3, όπου ορίζονται οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί των ενδιαφερομένων μερών, βλέπουμε ότι προβλέπονται οι καταναλωτές, οι εκπρόσωποι του περιβάλλοντος, οι κοινωνικοί εκπρόσωποι, οι μικρές και μεσές επιχειρήσεις, αλλά δεν υπάρχει βιομηχανία. Αναρωτιέμαι λοιπόν μήπως θα έπρεπε να τονίσουμε και την αντιγωνιστικότητα της βιομηχανίας μας μέσω αυτού του εγχειρήματο της τυποποίηση. και κάτι άλλο δευτερεύουν στον ε, ε, ε, ευρωπαϊκό Οργανισμό των Διαφερόμενων Μερών. Από ό,τι καταλαβαίνω, απαγορεύεται να υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων ε, με τι εμπορικέ, επαγγελματικέ πτυχέ ή άλλε. Αλλά μια οργάνωση, ένα ευρωπαϊκό οργανισμό που δεν έχει σύγκρουση συμφερόντων με τη βιομηχανία, το εμπόριο κτλ. είναι μια οργάνωση που κάνει πολιτική όλες οι οργανώσεις που γνωρίζουμε ουσιαστικά εκπροσωπούν αυτή την κατηγορία. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν πολύ καλά πώς μπορούμε να το διαθρώσουμε αυτό, κυρίως αν έχουμε ένα ευρωπαϊκό οργανισμό stakeholders που να έχει να κάνει με τη βιομηχανία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Η Επιτροπή μήπως θέλει να απαντήσει σε κάποιες από τις ερωτήσεις. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. να ξεκινήσω από τις τελευταίες παρατηρήσεις του κυρίου Οντί, γιατί είναι θέμα διευκρίνησης. Οι stakeholders, όπως τους αποκαλούμε, που αναφέρονται στο παράρτημα 3, είναι οργανώσεις που μπορούν να τύχουν χρηματοδότησης για τις δραστηριότητές τους στον τομέα της προτυποποίησης. Δηλαδή υπάρχει ένας κατάλογος αυτών των οργανώσεων που εκπροσωπούν κοινωνικά συμφέροντα ή μικρομεσαίων επιχειρήσεων και μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση. Η βιομηχανία, ο κλάδος αυτός καθεαυτός δεν θα λάβει χρηματοδότηση και γι' αυτό δεν αναφέρεται ο βιομηχανικός τομέας, δεν αναφέρεται καθαρά ο κλάδος στο παράδειγμα 3. Διαβάζοντας το διατακτικό του κανονισμού βλέπουμε ότι μπορούν να χρηματοδοτηθούν αυτοί οι τέσσερις μεγάλοι ευρωπαϊκοί οργανισμοί που εκπροσωπούν τα συμφέροντα της κοινωνίας ή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτούς μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε. Εδώ δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε ε, τον κλάδο. Βέβαια, οι εταιρείε του κλάδου βρίσκονται στην καρδιά της διαδικασίας προτυποποίησης, διότι διαμορφώνουν τα ευρωπαϊκά πρότυπα και αποτελούν ε, απαραίτητο εταίρο. Δεν μπορούμε να κάνουμε προτυποποίηση χωρίς τις εταιρείες του ίδιου του κλάδου. Και αυτό είναι βασικό στοιχείο για να καταλήξουμε σε πρότυπα που να μπορούν να γίνουν αποδεκτά από την αγορά. Τα πρότυπα αυτά πρέπει να έχουν διαμορφωθεί ε, στο πλαίσιο συνένεσης. Σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας στην προσέγγιση της Κομισιόν προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το ανέφερε και ο κύριος Μπιουτικόφερ. Όντως, προτείνουμε μια ισχυρότερη διατύπωση και ζητάμε από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης να εξασφαλίσουν την εκπροσώπηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Καταλαβαίνω την κριτική που μπορεί να υπάρξει για την διατύπωση αυτή, αλλά θεωρούμε, όπως και ο κ. Μπιτικόφερ και εσείς, πιστεύουμε ότι ασκούμε μια μεγαλύτερη πίεση, επιβάλλουμε μια μεγαλύτερη υποχρέωση και θα δούμε τι θα προκύψει από τη διαδικασία. Πάντως, όντως αυτό θέλουμε. Θέλουμε να δώσουμε πιο ισχυρό ρόλο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και δείχνει και τη δέσμευση που έχουμε αναλάβει προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και άλλους κοινωνικούς φορείς. Έχετε δίκιο ότι η συζήτηση γενικά θα στραφεί γύρω από τα βασικά σημεία του κανονισμού το ρόλο που θέλουμε να δώσουμε στι προδιαγραφέ τεχνολογία πληροφορική και επικοινωνιών και στον τομέα των υπηρεσιών. Για τον τομέα των υπηρεσιών, πολύ το ανέφεραν και ο κ. Μπιτικόφερ και ο εισήγητη, ότι δεν θα εφεύρουμε κάτι διαφορετικό για τι υπηρεσίε σε σχέση με αυτό που γίνεται για τα προϊόντα. Θα ακολουθήσουμε ακριβώ την ίδια διαδικασία για την κατάρτιση προτύπων. Θα βασιζόμαστε δηλαδή στις ανάγκες της αγορά την ίδια διαδικασία διαμόρφωσης προτύπων βάση συνένεσης. Δεν θέλουμε να επιβάλλουμε στον τομέα των υπηρεσιών κάτι που δεν θα αντικατοπτρίζει ε, τις επιθυμίες των ενδιαφερομένων. Αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε και στην ανακοίνωσή μας αλλά και στον κανονισμό. Στο πλαίσιο της σύνεσης που πολλοί παρεμβαίνοντες μας είπαν ότι είναι σημαντικό να επικρατεί. Για το τμήμα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών είναι η καρδιά του κανονισμού μας, γιατί αν θέλουμε ε, να συμβαδίζουμε με τις τεχνολογικές εξελίξεις, όπως έλεγε και ο κ. Μπιουτικόφερ, πρέπει να προσπαθήσουμε να επιταχύνουμε τους ρυθμούς, να χρησιμοποιήσουμε αυτά που ήδη υπάρχουν στην αγορά, άρα δεν πρόκειται να αρχίσουμε εμείς να διαμορφώνουμε πρότυπα, εφόσον ήδη Υπάρχουν πρότυπα που έχουν διαμορφωθεί από τα φόρουμ και συμπράξεις. Έχουμε ε, ορίσει κάποια σοβαρά ποιοτικά κριτήρια, κριτήρια που μας δίνουν όλες τις εγγυήσει. και δημιουργήσαμε και αυτή την πλατφόρμα που θα αποτελείται από όλου του ενδιαφερομένους στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Και κυβερνήσει, φόρουμ και συμπράξει, όχι οι επιχειρήσει αυτές καθεαυτέ. διότι όπως καταλαβαίνετε προσπαθούμε πάρα πολύ προσεκτικά να χειριζόμαστε τα θέματα που έχουν σχέση με ανταγωνισμό, πνευματική ιδιοκτησία κλπ. Βάζουμε κάποιες ρήτρες διασφάλισης, βάζουμε ε, ξεκινάμε μια διαδικασία για τον τομέα πληροφορικής και επικοινωνιών για να εγκρίνουμε προδιαγραφές που θα μας επιτρέψουν να υποστηρίζουν οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών πολύ σημαντικές πολιτικές μας, όπως είναι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονική υπογραφή κλπ. Χάρη σε αυτό το μηχανισμό λοιπόν προτυποποίησης στι τεχνολογίε πληροφορική και επικοινωνιών θα μπορέσουμε να προωθήσουμε πολλέ πολιτικέ μα. Αυτά προ το παρόν σε αυτό το πρώτο στάδιο ερωτήσεων. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μία ερώτηση προς τον κύριο Γκίρεκ, προς τον εισηγητή. Θέλετε εσείς κύριε Γκίρεκ να ξαναμιλήσετε ή είστε ικανοποιημένος με τα όσα έχουν λεχθεί μέχρι τώρα. Ευχαριστώ. Να αντιδράσω για δύο θέματα. Καταρχήν ε, για τον ε, ορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και των προτύπων. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει οι ορισμοί αυτοί να είναι πολύ σαφείς σύμφωνα με τα πρότυπα ISO. Γιατί αυτά είναι τα πρότυπα που ε, κάνουν τη διαφοροποίηση μεταξύ προδιαγραφών και προτύπων ε, και εδώ συμφωνώ με τον συνάδελφο για το θέμα αυτό. Για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να πω το εξή. Φυσικά και πρέπει να συμμετέχουν ε, στη δημιουργία εκπόνησης προτύπων και προδιαγραφών, αλλά πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία εκπόνησης λοιπόν, αλλά πρέπει να σέβονται συγκεκριμένους ε, κανόνες. Γι' αυτό έχω αυτή την τροπολογία υπαριθμών 18 και λέω facilitating ε, και όχι ensure, γιατί όρου ensure διασφαλίζω. Σημαίνει ότι θα πληρώνουν για τη συμμετοχή τους. Δεν ξέρω αν ε, οι οργανισμοί προτύπων ε, είναι έτοιμοι να συνεισφέρουν τον τρόπο αυτό για την εμπλοκή των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Κατά τα λοιπά, συμφωνώ με τους ομιλητές που είπαν ότι πρέπει να υπογραμμίσουμε τη σημασία των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και να προωθήσουμε το ρόλο τους ε, στην εκπόνηση προτύπων και τεχνικών προδιαγραφών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Γκύρε και ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους και την Επιτροπή. Και κλείνουμε αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης. Προθεσμία για την κατάσταση τροπολογιών 12 Ιανουαρίου. Δεν υπάρχουν αντιρρήσει. Κλείνει λοιπόν αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης. Κάνουμε 5 λεπτά διάλειμμα και να είμαστε εδώ στις 10 για τις ψηφοφορίες. Σύντομο διάλειμμα.

Κυρίε Κυρίες και κύριοι, ας ξεκινήσουμε. Δεν ξέρω γιατί, αλλά μου φαίνεται ότι είμαστε λιγότερο πολυπληθεί σήμερα. Μάλλον θα έχει σχέση με το ότι κοντεύουμε προς το τέλος της εβδομάδας. Ελπίζω το απόγευμα να είμαστε πολυπληθέστατοι γιατί θα έχουμε και εκπρόσωπο της Προεδρίας και δεν θα φαίνεται ωραία να είμαι εγώ μόνος μου εδώ. Ελπίζω λοιπόν το απόγευμα να είναι εδώ πολλοί συνάδελφοι. Ας ξεκινήσουμε με την έκθεση της κυρίας Λένα Κολάσκα Μπομπίνσκα. Ε, ζητώ συγγνώμη εκ μέρους της διότι δεν μπορούσε σήμερα να είναι παρούσα. Έχει κάποιο οικογενειακό πρόβλημα. Μπορούμε να ξεκινήσουμε όμως χωρίς την κυρία Κολάσκα Μπομπίνσκα. Ξεκινάμε λοιπόν. Έχετε όλες τις κάρτες ε, ε, για, να ελέγχουμε την ψηφοφορία. Τι θα κάνουμε. Ξεκινάμε. Συμβαστική τροπολογία 1. Όχι, όχι, όχι, όχι. όχι. Ήδη ξεκινάμε καλά. Charles. Ζητώ την επίοικιά σας, Πρόεδρε δεν έχει κάρτα ψηφοφορία η συναδελφό μου. Α γίνει λοιπόν διανατάσσεως τη χειρό. Ζητώ συγγνώμη, μάλλον δικό μου λάθο θα είναι. Okay. Also, es fehlt eine Karte. Λοιπόν, λείπει μία κάρτα. Ε, δεν φαίνεται να είναι και τόσο δραματικά. Τούρμε ούτε εσείς κάρτα. Και, μη, και κάποιος από εμά δεν έχει κάρτα, πρέπει να το δούμε. Λοιπόν, μία κάρτα λείπει από το ECR και άλλη μία από, το, από τους πρασίνους. Όλες οι άλλες ομάδες έχουν όλες τις κάρτες. Πολύ ωραία. Ξεκινάμε. Συμβαστική τροπολογία Α. Ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, αποφασίζεται. Τροπολογία Β. Κατά, αποχές, αποσύρεται. Συμβαστική τροπολογία Γ, σε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία Δ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Περνάμε στο 9, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 10, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 11, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 14. Καταπίπτει. Σωστά. Όχι. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 15 καταπίπτει. Συμβαστική τροπολογία ε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Καταπίπτουν όλα τα υπόλοιπα. 26.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 Ωραία. Λοιπόν, πέραση τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 41 ψήφοι υπέρ. Απορρίπτεται. 41. 42 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 43 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Περνάμε στη συνολική ψηφοφορία με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Στο ΕΛΚ έχουμε έναν παραπάνω. Zwei? Zwei zu Πέρας της ψηφοφορίας. Συγχαρητήρια. Τι, συν ένα, συν δύο, συν δύο, συν δύο. Κατά. Α, ένας υπέρ, ένας κατά. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Και περνάμε στην έκθεση Γκλάντε, που και εκείνο δεν είναι εδώ γιατί είναι άρρωστος. Περαστικά του. Πήγα να πω χρόνια πολλά, ε, περαστικά εννοούσα, τι άλλο δεν εννοούσα. Θα του τα μεταφέρουμε. Λοιπόν, ψηφοφορία. Έχουμε ένα κείμενο συμβιβαστικό. Ποιο ψηφίζει υπέρ του συμβιβαστικού κειμένου. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται και περνάμε στην τελική ψηφοφορία. Με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Αυτή τη φορά δεν έχουμε παραπανήσει ψήφους. Πέρασε τη ψηφοφορία. 42 και άλλοι δύο συν 44. Με τεράστια πλειοψηφία θα του το στείλουμε σαν δωράκι για το χριστουγεννιάτικο δένδρο. Τελειώσαμε λοιπόν με τις ψηφοφορίες. Και μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο της της διάταξης, εφόσον συμφωνείτε, που είναι το περίφημο σημείο ενεργειακή απόδοση. Συνάδελφος Τούρμες έχει το λόγο. Φαντάζομαι ότι έχετε όλο το πακέτο. Το πήρατε όλο το πακέτο? Έχουμε ένα βουνό από τροπολογίες. Θα σας βοηθήσει η γραμματεία αν δεν μπορείτε να τα κουβαλήσετε. Κλοντ, θες να ξεκινήσεις? Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πριν αρχίσει ο Κλοντ, να θέσω εγώ ένα θέμα. Συγκεκριμένα, χρονοδιάγραμμα για αυτό το φάκελο. Νομίζω ότι και εσείς είπατε πολύ σωστά ότι είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός των τροπολογιών. Ελπίζω λοιπόν να μην προσπαθήσουμε να βιαστούμε. Καλύτερα να παραταθεί η προθεσμία παρά να προσπαθήσουμε να το κάνουμε βιαστικά και γρήγορα. Αυτή είναι η παράκλησή μου προς τον εισηγητή και τους Κιώδης, διότι πρόκειται για σημαντικό νομοθέτημα. Νομίζω και ελπίζω ότι μπορούμε να είμαστε ευέλικτοι ως προς το χρονοδιάγραμμα. Ευχαριστώ. Ωραία, ο Κλόντ είναι ο επόμενο Αγαπητοί συνάδελφοι, θα είμαι πάρα πολύ σύντομο ε, στην εισαγωγή μου. Πρώτον, σε ό,τι αφορά τη διαδικασία. Φυσικά, έχετε δίκιο, είναι πρόκληση να αντιμετωπίσουμε τις 800 και τροπολογίες, αλλά χάρη ε, στο προσωπικό της γραμματείας ε, των ομάδων μας ε, και στις προσπάθειες των σκιωδών Κάναμε μια σειρά συναντήσεων και διαπραγματεύσεων και έχουμε προβλέψει πέντε συναντήσεις ακόμη ε, με τους σκιώδεις. Θα έχουμε και ε, απόψε το απόγευμα άλλη μια συνάντηση για να δούμε αν είμαστε στο δρόμο που έχουμε χαράξει ακόμη. Και αν δούμε ότι είναι εντελώς αδύνατο να έχουμε τέλη Ιανουαρίου μια ψηφοφορία, θα το συζητήσουμε του χειώδεις, ίσως το μεσημέρι, το απόγευμα σήμερα και θα δούμε που θα καταλήξουμε. Για να καταλάβετε λίγο πολύ τι γίνεται, μετά την σημερινή συνεδρίαση θα έχουμε δει ίσως ε, διεκπαιρεώσει αρκετές από τις 800 τροπολογίες, 150-200, Ελπίζουμε να μην έχουν μείνει πάρα πολλές. Αυτά σε ό,τι αφορά την διαδικασία. 1.100-1.200 τροπολογίες περίπου θα τις έχουμε διεκπαιρεώσει. Γιατί λοιπόν τις κυβερνήσεις, επιχειρήσεις ε, και εμάς, γιατί μας ταλαιπωρούμε με αυτό το νομοθέτημα. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στην Ευρώπη. Περί αυτού πρόκειται λοιπόν. Και θα σας δώσω τρία σύντομα παραδείγματα. Η οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το εμπορικό ισοζύγιο πληρωμών το 2009 είχαμε ένα μικρό έλλειμμα, γύρω στα 4 δις. Το 2010 είχαμε θετικό πρόσημο, γύρω στα 10 δις ήταν το πλεόνασμα. Γιατί το λέω αυτό. Για να καταλάβουμε ότι δαπανούμε κάθε χρόνο 400 δις περίπου για την αγορά πετρελαίου και φυσικού αερίου. Αυτό σημαίνει ότι τη Ρωσία, την Νορβηγία, τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ ε, βοηθάμε να πλουτίσουν. Μεταφέρουμε γιατί η ενέργεια ουσιαστικά είναι μια μεταφορά πλούτου από τις ευρωπαϊκές οικονομίες σε άλλες οικονομίες του κόσμου. Ο στόχος μου, αυτός ο στόχος του 20% ουσιαστικά έχει να κάνει με την μείωση αυτής της μεταφοράς πλούτου. 400 δις που μεταφέρονται, ας μειώσουμε κατά 50 δις ή λίγο παραπάνω τη μεταφορά πλούτου στις οικονομίες τρίτων χωρών. Η ενεργειακή απόδοση τριτων χωρων ενεργειακη επενδύσεις με αυτό πολλές φορές έχουν να κάνουν με τοπικές ε, θέσεις εργασίες. Τοπικέ λοιπόν δουλειέ δεν έχουμε ανταγωνισμό με την Κίνα παραδείγματο χάρη με την κινέζικη οικονομία. Και επίση η τεχνολογία σε πολύ μεγάλο βαθμό ε, παράγεται εδώ, στην Ευρώπη. Άλλο είναι αυτό, η ενεργειακή απόδοση και άλλο οι επίπεδε οθόνε, τα flat screen στην τηλεόραση που τα εισάγουν σχεδόν 100% τα προϊόντα αυτά. Μπορούμε λοιπόν να κάνουμε τη διαφορά. Ένα δεύτερο θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό ανταγωνιστικότητα έντασης ενέργειας, ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τι προσπαθούμε να πετύχουμε με την οδηγία αυτή. Ουσιαστικά προσπαθούμε να μειώσουμε το κόστος ε, για την ενέργεια της μικρομεσαίας επιχειρήσης. Πώς μπορούμε να το μειώσουμε το κόστος, μπορούμε να μειώσουμε τον όγκο. Μπορούμε να βοηθήσουμε την έρευνα για την ενέργεια, ε, για βελτίωση των διαδικασιών παραγωγής ε, και μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση. Πρέπει όμως να καταλάβουμε το εξής. Έχουμε απελευθερώσει τις ε, αγορές ηλεκτρισμού. Η τιμή λοιπόν βασίζεται στο πιο, στην πιο υψηλή ε, στο πιο ψηλό τιμολόγιο, στο πιο ψηλό ε, στην πιο ψηλή τιμή σε μια μονάδα παραγωγής ενέργειας. Πρέπει να δούμε όμως και την καμπύλη. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τις τιμές να εξελιχθούν στην ε, Λιψία, στη Μαδρίτη, στο Άμστερντο, στο Παρίσι η τιμή του ρεύματος ίσως να μπορούσε να πέσει. Στις αγορές εκεί όπου αγοράζει κανείς ρεύμα ουσιαστικά. Και στρέφουμε προς την Κομισιόν. Όταν εξετάσετε τις λεπτομέρειες της οδηγίας θα δείτε ότι αποκλείεται η μη χρήση ενέργειας από τη μοντελοποίηση και από τους στόχους. Δηλαδή, τελικά έχω δίκιο αν πω ότι ο άνθρακας που θα μπει σε μία ψυκάμινο δεν λαμβάνεται υπόψη ή διαδικασίες ε, χημικής ε, μετατροπής δεν λαμβάνονται υπόψη. θα μπορούσε να μας εξηγήσει η Κομισιόν. Ο αυτός ο αποκλεισμός, αυτή η εξαίρεση της μη χρήσης ενέργειας, non-energy use. Την προηγούμενη εβδομάδα μας παρουσίασε επίσης ε, ένα οδικό χάρτη Κομισιόν. Λέει, πυρηνικό, πυρηνική, άνθρακα, ανανεώσιμες μειώνονται. Λόγω του κόστους του ηλεκτρισμού όμως θα αυξηθεί η, ενέργεια, η τιμή της ενέργειας γιατί τα παλιά εργοστάσια πρέπει να αντικατασταθούν και οι παλιές γραμμές παροχής ισχύω πρέπει να αντικατασταθούν. Στον οδικό χάρτη λοιπόν το ποσοστό των δαπανών των ευρωπαϊκών νοικοκυριών θα αυξηθεί σε ό,τι αφορά το ενεργειακό κόστος. Άρα και με αυτή την νομοθεσία μπορούμε να βοηθήσουμε ιδίω τα νοικοκυριά τα οποία ενεργειακά μπορούν να χαρακτηριστούν ως φτωχά. Μπορούμε, μπορούμε πιστεύουμε να βοηθήσουμε με την οδηγία αυτή και προς αυτή την κατεύθυνση. Ε, σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα για τη διαδικασία, για να μην κάνουμε κανένα λάθος. Ο εισηγητή και οι σκιώδεις εισηγητέ μας βοηθούν πολύ και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας βοηθάτε με τις συμβιβαστικές τροπολογίες, αλλά το χρονοδιάγραμμα μόνο η Επιτροπή μπορεί να το αποφασίσει, δεν μπορεί να το αποφασίσει κανείς άλλος σε, στενότερο κύκλο. Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα μέχρι ότου το αποφασίσουμε. Κανένα χρονοδιάγραμμα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Απλώς θα πρέπει να συμφωνήσουμε, επιθυμία όλων μας είναι αυτό, να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε κάπως και ελπίζω με την Δανέζικη Προεδρία να έχει ολοκληρωθεί το θέμα. Αυτό είναι η επιθυμία μας. Μπορεί να χρειαστεί να αναβάλουμε την ψηφοφορία μια-δυο εβδομάδε. Δεν υπάρχει πρόβλημα από αυτού σε σχέση με τα σχόλια που έκαναν οι προηγούμενοι ομιλητέ. Θα έχουμε την ισχύ και τον Ιανουάριο να το εξετάσουμε. Πάντω είναι αρκετά πολύπλοκο το θέμα, πολλά σημεία. Έχω αρκετού ομιλητέ Α, πρέπει να ξεκινήσουμε με τους σκιώδεις. Λοιπόν, ο κύριος Πίπερ είναι πρώτος, μετά η κυρία Τόνση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι επενδύσεις στην αποδοτικότητα της ενέργειας ε, είναι θέματα ιδιαίτερα ε, σημαντικά και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε και για λόγους κόστους, για να χρησιμοποιείται λιγότερη ενέργεια και για να μειώσουμε την εξάρτησή μας από την ενέργεια, όπως πολύ σωστά είπε ο συνάδελφος ε, Τούρμες. Ο κύριος Τούρμες όμως δεν είπε αυτά τα οποία έχουμε στη μείσια διάταξη για σήμερα που πρέπει να μιλήσουμε για τις τροπολογίες. Θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα θετικά σημεία. Έχουμε κάποια μικρά βήματα τα οποία πρέπει να κάνουμε μαζί στο άρθρο 2 για τις δυνατότητες χρηματοδότησης παραδείγματος χάρη για την ενεργειακή απόδοση και στο άρθρο 10 για τη συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας και εδώ βλέπω κάποια δυνατότητα να συμφωνήσουμε αλλά σε βασικά ζητήματα δίστανται κατά πολύ οι απόψεις μας. Ο εισηγητής εδώ τονίζει πάρα πολύ κάποιες λεπτομέρειες. Εμείς θέλουμε μια γενική δέσμευση των κρατών μελών για την ενεργειακή απόδοση και μετά οι πολίτες, οι επιχειρήσεις και τα κράτη-μέλη να έχουν μια μεγαλύτερη ευελιξία για το πώς θα επιτύχουν τους στόχους. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η τακτική του εισηγητού οι συμβιβαστικές, οι συμβιβασμοί δεν είναι συμβιβασμοί, κύριε Τούρμες. Έχετε κάποιες ε, τροπολογίες με 10% με 20% που είναι όλες προς τη δική σας κατεύθυνση όμως. Δηλαδή εντείνουν ε, τη δική σας ε, προσέγγιση αυτά τα οποία έχετε αποδεχθεί. Δεν έχετε κάνει καμία κίνηση προς τις άλλες κατευθύνσεις. Και δυστυχώς υπάρχουν ακόμη αρκετά ανοιχτά θέματα. Στο άρθρο 3, εκεί όπου λέμε ότι μέχρι το 2050 θέλουμε μία μείωση κατανάλωση για όλα τα κτίρια και υπάρχει μάλιστα και ένας δεσμευτικός στόχος 80%. Δεσμευτικός στόχος 80% για τα κτίρια, κύριε Τούρμες χρόνια πολλά και για τα γενέθλιά σας που μόλις πέρασαν. Το 2050 θα είστε 91 ετών. Και, και εγώ 89. Εσείς είστε πιο, σε πιο καλή φυσική κατάσταση από μένα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, στα 80 και στα 90 μας ακόμη αυτή την πολιτική θα συζητάμε. Ε, ε, ε, τι είναι αυτό το οποίο τώρα συζητάμε. Μιλάμε για επενδύσεις για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, για τις αγορές. Δεν μπορούμε σήμερα να βάλουμε δεσμευτικούς στόχους για 30 και 40 χρόνια αργότερα. Εδώ μιλάμε για το στόχο εξοικονόμησης ενέργειας για το 2020, κάτι το οποίο πρέπει το συντομότερο δυνατόν να επιτύχουμε. Τώρα τα υπόλοιπα για 40 χρόνια αργότερα είναι κάτι σαν επιστημονική φαντασία. Θα έχουμε να τα συζητήσουμε πολλά χρόνια. Και θέλω να πω και κάτι ακόμη το οποίο και τώρα συζητείτε και ψηφίζετε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος για το σύστημα ε, εμπορίας εκπομπών ε, διοξιδίου του άνθρακος και τα σχετικά πιστοποιητικά. Έχουν γίνει πολύ φτηνά αυτά τα πιστοποιητικά. Αυτές οι άδειε για ε, το διοξιδίου του άνθρακος έχουν γίνει πάρα πολύ φτηνές. Τι θα πρέπει να κάνουμε λοιπόν. Υπάρχουν προτάσεις τις οποίες διαβάζουμε και μας εκπλήσουν και εδώ νομίζω ότι θα πρέπει να αφήσουμε το θέμα των εκπομπών ε, διοξιδίου του άνθρακος και θα πρέπει και η Επιτροπή να αξιολογήσει τα θέματα της εμπορίας, του συστήματος εμπορίας εκπομπών. Μια και μιλάμε για τις τροπολογίες, θα ήθελα να μιλήσω και για τα συγκεκριμένα άρθρα. Στο άρθρο 3 έχουμε το στόχο του 20% κάτι το οποίο εμείς ως ΕΛΚ αναγνωρίζουμε και δεσμευτικά, αλλά θα πρέπει να αφήσουμε ελευθερία επιλογής για τα κράτη-μέλη. Ορίζουμε στόχους για την παραγωγικότητα στην ενέργεια και σε συγκεκριμένους τομείς μέσα στην ε, ε, παραγωγικότητα για την ενέργεια. Υπάρχει ο συνολικός στόχος, αυτός δεν αμφισβητείται, αλλά μιλάμε για την ευελιξία που πρέπει να αφήσουμε στα κράτη-μέλη να δράσουν κατά τον καλύτερο τρόπο ώστε να επιτύχουν αυτό το στόχο. Ε, τέταρτο άρθρο για την ανακαίνιση κτηρίων. 3% ε, της επιφάνειας ε, ανακαίνιση ετησίως. Από πολλές χώρες θεωρείται αυτό ουτοπία. Άλλοι βέβαια λένε ότι έχουμε προχωρήσει και περισσότερο. Και εδώ πάλι χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία να σκεφτούμε και τους ενοικιαστές, να σκεφτούμε και τις κοινωνικές ε, απαιτήσει. Δεν μπορούμε να το ορίσουμε καθοριστικά και δεσμευτικά για όλους. Μέχρι το 2018 θα πρέπει ε, να έχουμε κατοικίες ε, με χαμηλή ενέργεια και όταν ενοικιάζονται κάποια κτίρια θα πρέπει να έχουν τη χαμηλότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας. Αυτό θα μπορούσε να ισχύσει και για τα δημόσια κτίρια ε, ε, τα οποία νοικιάζουμε εδώ στις αντιπροσωπείες μας, στις αντιπροσωπείες των κρατηδίων της Γερμανίας. Έτσι και, βάλουμε, έτσι και επιβάλλουμε τέτοια υποχρέωση. Νομίζω ότι ε, όλοι θα, θα εκπλαγούν. Ας λίγο πιο ρεαλιστικοί με τις ε, τροπολογίες, με τις ε, προτάσεις μας. Ίσως στον ιδιωτικό τομέα κάποιος να θέλει να επιτύχει ε, κάτι περισσότερο και να τα καταφέρνει. Ίσως ε, και στο δημόσιο τομέα να ε, επιτευχθούν πρόοδοι. Αλλά ας αφήσουμε λίγο μεγαλύτερη ευελιξία και στα κρατημέλη και σε όλους για να μπορέσουν για την ανακαίνιση κτίριων να κάνουν τα βήματα με τον καλύτερο δυνατό ρυθμό. Στο άρθρο 5, σχετικά με τις προσκλήσεις υποβολής ενδιαφέροντος και το δημόσιο τομέα, λέτε ότι η αποτελεσματικότητα της ενέργειας είναι πολύ σημαντική σε μια πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος, εξίσου σημαντική με την τιμή, με το τίμημα της σύμβασης. Ε, υπάρχουν διάφορα πολύ σημαντικά. Υπάρχει η συμμετοχή των γυναικών, υπάρχει η κοινωνική συμμετοχή των επιχειρήσεων δεν μπορούμε να αφαιρούμε τα δικαιώματα από τους Δήμους, από τις κοινότητες. Ε, ε, μπορεί το επόμενο που θα μας προτείνετε να, να, είναι αυτό. Αν τώρα επιτύχουμε αυτό, το επόμενο βήμα θα είναι ε, να πάρουμε κάθε δικαίωμα και από τους Δήμους και κοινότητες. Δεν είναι αιτιολογημένα λοιπόν αυτά τα οποία προτείνονται. Στο άρθρο 6 τώρα. Και εδώ θέλουμε εξοικονόμηση 1,5% συμφωνούμε αλλά και εδώ πάλι δεν μπορούμε όλα να τα αποφασίσουμε με τον ίδιο τρόπο. Πρέπει να μπορούν τα κράτη-μέλη μόνο τους να αποφασίζουν ε, την οδό που θα ακολουθήσουν. Θέλουμε βελτίωση των ε, σταθμών παραγωγής ε, ενέργειας και βελτίωση στις μεταφορές. Πολύ συχνά υπάρχουν και μακροπρόθεσμα μέτρα όταν αλλάζουμε μία ε, ε, ηλεκτρική συσκευή, παραδείγματο χάρη, θα πρέπει και εκεί να υπάρχει δυνατότητα ε, πρόοδου και εξοικονόμηση. Υπάρχουν και μακρο... βραχυπρόθεσμα μέτρα τα οποία θα έπρεπε ο κ. Τούρμες να αναγνωρίσει για την έξυπνη παροχή. Επίσης θα έπρεπε να προβλέπουμε κάτι. Δεν μπορούμε να έχουμε μόνο συσκευέ ε, σε μια αγορά λιγότερο από 3%. Οι μετρήσει πώς θα γίνονται, από ποιον και πότε. Και θα σας δώσω και ένα παράδειγμα ε, ε, ε, και πολλά παραδείγματα για να σας εξηγήσω πόσο περίεργα είναι όλα αυτά. Όταν αγοράζουμε ένα ψυγείο που είναι α με τρία συν, που σημαίνει ότι είναι υψηλής ενεργειακής απόδοσης, εξοικονομεί ενέργεια και εμείς δαπανούμε λίγα χρήματα για την ενέργεια. Αν πολύτε ένα ψυγείο με συντελεστή C, με μέτρηση C, τι εξοικονόμηση υπάρχει. θα πρέπει να υπάρχει και κάποιος τρόπος μέτρησης για να μπορούν τα κράτη-μέλη να αξιολογούν την πρόοδο που έχουν κάνει μέχρι κάθε ε, δεδομένο σημείο. Και υπάρχει και το φαινόμενο rebound όπως ονομάζεται. Όταν αγοράζουμε ε, ένα ψυγείο και το βάλουμε στο υπόγειο γιατί θέλουμε να βάλουμε τις μπύρες μας να κρυώνουν στο υπόγειο, τι θα αποφασίσουμε. Θα, θα πάρουμε εμεί αποφάσει για μια οικογένεια που βάζει τις μπύρες στο υπόγειο σε ένα νησί του Αιγαίου ή στη Λιθουανία δεν μπορούμε εμείς να προσδιορίσουμε τι ακριβώς θα κάνει ο κάθε πολίτης. Και το παράρτημα 5 ε, ε, πιστεύω πραγματικά δεν είναι δυνατόν ε, να το θεωρούμε λογικό. Εξετάστε το λίγο προσεκτικότερα. Για την ενεργειακή αποδοτικότητα είπαμε ότι συμφωνούμε, θέλουμε να έχουμε στόχους, θέλουμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα και θα πρέπει να συμφωνήσουμε και για τα μέτρα. Τα μέτρα που θα χρησιμοποιήσουμε θα πρέπει να είναι ευέλικτα. Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει δικαίωμα παρέμβασης και τα κράτη-μέλη να, να μπορεί να τα επαναφέρει στο σωστό δρόμο. Νομίζω ότι θα, μπορέσουμε, θα καταφέρουμε να δημιουργήσουμε ταραχή στα κράτη-μέλη αν επιμείνουμε με δεσμευτικά μέσα περισσότερο όπως πρέπει. Ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφος Τόμσον. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ όλους για όλη τη συνεισφορά σας και για την υποβολή τόσο πολλών τροπολογιών όπως ακούσαμε από τον κύριο Τουρμές πάνω από 800 τροπολογίε και 300 τροπολογίε μόνο για το άρθρο 10. Αν ε, έτσι λοιπόν ε, και η γραμματεία και ο εισηγητής ε, αλλά και το προσωπικό έχουν το δύσκολο έργο να βρουν συμβιβασμούς. Όπως ακούσαμε είναι πάρα πολύ δύσκολο αλλά εργαζόμαστε σκληρά για να καταλήξουμε σε συμφωνία. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους λοιπόν και τον Κλοντ για την πολύ καλή δουλειά που υλοποιεί αυτή τη στιγμή. Για πολύ καιρό ακούσαμε τους καταναλωτές, ε, τη βιομηχανία, τα συνδικάτα, τις ε, διάφορες οργανώσεις ε, και φυσικά και τους συναδέλφους στην Επιτροπή Ήτρε και εγώ εκ μέρους της ομάδας των σοσιαλιστών βρήκα ότι λείπουν κάποια, πράγματα από την πρόταση της Κομισιόν αλλά πριν το πω αυτό θέλω να απαντήσω στον κύριο Πίπερ σε σχέση με τις μακροπρόθεσμες ε, προοπτικές. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή τη μακροπρόθεσμη προοπτική 2050. Στην οδηγία αυτή, όπως ε, και σε όλες τις άλλες οδηγίες, εδώ μιλάμε για χάραξη πολιτικής. Εδώ και τώρα και αν κάνουμε πολιτική χωρίς προοπτική, αυτό μας οδηγεί σε κρίση στην Ευρώπη. Έτσι λοιπόν σας ευχαριστούμε για αυτή την προοπτική μέχρι το 2050. Πέραν αυτού. Νομίζω ότι αυτό που χρειαζόμαστε είναι ο δεσμευτικός στόχος. Ε, φυσικά θα πρέπει να υπάρχει ευελιξία, αλλά 20% ενεργειακή αποδοτικότητα δεν είναι κάτι καινούριο. Το αποφασίσαμε αυτό και στο Συμβούλιο, όταν η κυρία Μέρκελ ήταν πρόεδρος του Συμβουλίου, αποφάσισε 20% ενεργειακή αποδοτικότητα και ε, ψηφίσαμε το Δεκέμβριο του 2008 σε αυτό το κοινοβούλιο για την οδηγία για τις ανανεώσιμες 20% ενεργειακή αποδοτικότητα. Δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε λοιπόν το αν είμαστε υπέρ ή όχι της ενεργικής αποδοτικότητας. Το πρόβλημα είναι ότι ήμασταν πάρα πολύ ευγενικά, ευγενικοί στα κρατημέλη και δεν είπαμε δεσμευτικό στόχο. Και τι κάνει το κρατημέλη, δεν κάνουν τίποτα, τίποτα απολύτω. Και έτσι λοιπόν πρέπει να του πούμε, πρέπει να έχετε δεσμευτικού στόχου φυσικά, γιατί Διαφορετικά είναι πολύ κακό το μήνυμα και γιατί πρέπει να στείλουμε μήνυμα δεσμευτικού στόχου, όπως είπε η Αγίλα Μέρκελ, Πρόκειται για ένα μήνυμα στην ε, βιομηχανία, στον κλάδο. Γιατί ποιος θα επενδύσει σε κάτι που δεν είναι δεσμευτικό στόχος. Άκουσα τι προάλλε ε, ότι στη χώρα μου τα εξοδοξικά ταμεία ε, έχουν πάρα πολλά χρήματα και δεν ξέρουν πού να τα επενδύσουν. Θέλουμε να επενδύσουν ε, δηλαδή στην ε, ενεργειακή αποδοτικότητα, αλλά δεν υπάρχουν δεσμευτικοί στόχοι, δεν υπάρχουν εγγύησει, δεν τολμούν να επενδύσουν εκεί. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό. Να κάνουμε τα κράτη-μέλη να κατανοήσουν ε, τα χρηματοδοτικά μέσα και να προωθήσουμε τη δημιουργία αγορών ΕΣΚΟ, εταιριών εξοικονόμησης ενέργειας, έτσι ώστε να εφαρμοστούν σωστά τα 4 και 6. Τα κράτη-μέλη λοιπόν θα πρέπει να θέσουν ε, μία σειρά μέσων χρηματοδότησης ε, τώρα για την ομάδα σοσιαλιστών και δημοκρατών. Εμείς ε, θεωρούμε και το θέμα της ανέχειας πάρα πολύ σημαντικό και το θέμα της κατάρτισης, γιατί δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε όλες αυτές τις φανταστικές θέσεις εργασίας σε τοπικό επίπεδο που θα δημιουργηθούν με αυτή την οδηγία χωρίς ε, να ξεκινήσουμε μια διαδικασία κατάρτισης στην Ευρώπη γιατί δεν έχουμε τώρα τις ικανότητες. Άρθρο 6 και άρθρο 12. Λένε και τα δύο ότι ο κοινωνικό στόχο μπορεί να είναι τμήμα των συστημάτων ε, της εξοικονόμηση ενέργειας. Πρέπει να τονίσουμε αυτή τη διατύπωση και να την καταστήσουμε το το ΣΑΛΠ. αλλά πολλοί από τους συναδέλφους και οδείς ανησυχούν για την ευελιξία ε, για τα κράτη-μέλη και τις εταιρείες παρά να ε, την ανέχεια στον τομέα της ενέργειας. Θα μπορούσε βέβαια αυτό να είναι τμήμα και των εφιών, της εφιούς μέτρησης Όμω μπορεί να μην είναι και τόσο ευφύ όσο ακούγεται. Μου αρέσει η ιδέα οι καταναλωτέ να μπορούν να βλέπουν και να αντιδρούν σε πραγματικό χρόνο στην ενεργειακή δημολόγηση, Αλλά αυτό δεν είναι ακόμα δυνατόν και δεν θα πρέπει να ε, αναγκάσουμε τα κράτη-μέλη να αποκλείσουν του έξυπνου μετρητέ. Ε, έξυπνοι μετρητέ, επίση μετρητέ, τι σημαίνει ότι μπορείτε να ε, καταναλώσετε ενέργεια όταν είναι φτηνή. Το 2006 με προσκάλεσαν ε, να μιλήσω στη Σόφια σε ένα συνέδριο για τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια ε, που οργανώθηκε από το Γερμανικό Ίδρυμα Βάιμπουργκ. Πήγα εκεί και ε, βοηθός του διευθυντή μου είπε είμαι τόσο κουρασμένη, δεν κοιμήθηκα χθες το βράδυ και είπα γιατί δεν κοιμήθηκες. Και μου είπε εδώ στη Βουλγαρία είναι πιο φθηνή ενέργεια μετά ε, τα μεσάνυχτα έτσι λοιπόν, οι φτωχοί άνθρωποι εγώ, γιατί είμαι μόνη μητέρα, μαγειρεύουμε ε, και πλένουμε κατά τη διάρκεια τη νύχτα. Έτσι λοιπόν δεν προλαβαίνουμε να κοιμηθούμε. Έτσι λοιπόν, ε, αν έχουμε τσιβεί μετρητές, ε, ε δεν ε, θα λύσουμε απαραίτητα το πρόβλημα της ενεργειακής ανέχειας. Χρειαζόμαστε μια φιλόδοξη οδηγία για την ενεργειακή αποδοτικότητα, όχι γιατί είναι κάτι που μας βολεύει, αλλά επειδή είναι απαραίτητη και είναι αποτελεσματική προς ως προς το κόστος. Είναι σημαντικό και για την Προεδρία της Δανίας, μας είπαν. Μπορώ να σας πω ότι η οδηγία για την ενεργειακή αποδοτικότητα είναι πράγματι πάρα πολύ σημαντική για την Προεδρία της Δανίας, όχι μόνο γιατί έχουμε αυτή την πολύ καλή εμπειρία με την εξοικονόμηση ενέργειας στη Δανία, στο τέλη του 70, στις του 70, ως ε, απάντηση στην παγκόσμια πετρελαϊκή κρίση, δύο χώρες αντέδρασαν, η Βραζιλία αντέδρασε με την ε, δημιουργία του συστήματος βιοκαυσίμων και η Δανία με τη δημιουργία του σχεδίου θέρμασης της Δανίας, δηλαδή για 20 ε, χρόνια δεν έχει αυξηθεί η κατανάλωση ενέργειας στη Δανία, ενώ η οικονομία αυξήθηκε, η κατανάλωση της ε, μεγενθήθηκε, με συγχωρείτε, η κατανάλωση ενέργειας δεν αυξήθηκε στη Δανία. Έτσι λοιπόν ε, θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας αυτή την εμπειρία και νομίζω ότι μπορείτε να μάθετε πολλά από το παράδειγμα της Δανίας, αλλά φυσικά κάθε χρόνο βάζουμε 200 δισεκατομμύρια ευρώ στις ε, τσέπες του Πούτιν. Το 50% ε, της ενέργειας στην Ευρώπη ε, εξάγεται σε εμά ε, και οι μισές εξαγωγές προέρχονται από τη Ρωσία. Έτσι λοιπόν αυτά τα χρήματα πηγαίνουν στις τσέπες του Πούτιν, χρήματα που θα μπορούσαμε να έχουμε ξεκονομήσει και να επενδύσουμε σε εργασίες στην Ευρώπη, σε τοπικό επίπεδο όπως είπε ο κ. Στούρμας πριν. το χάρη μόνωση των κτηρίων στην Ευρώπη δεν μπορεί να τεθεί στους Κινέζους. Έτσι λοιπόν, πολλά μπορούμε να πούμε για την ενεργειακή αποδοτικότητα, για την οδηγία, της διαπραγματεύσεις και τις τροπολογίες, αλλά δεν θα μακρηγορήσω εγώ περισσότερο. Θα τα πω καλύτερα στη συνάντηση του Σκιωδών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Συνάδελφο Φόρντ είναι η επόμενη μιλητία. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τους συνεργάτες του που κάνουν ε, πάρα πολύ δουλειά γιατί είναι πραγματικά δύσκολο ε, να συμπληρώσει κανείς διαφορετικές απόψεις και τόσο πολλές τροπολογίες. Σας έφερα από τη χριστουγεννιάτικη αγορά κύριε Τούρμε σε ένα δωράκι χριστουγεννιάτικο έτσι να σε δωροδοκίσω λίγο να λάβεις υπόψη σου τις απόψεις μας. Um, Obviously, you know... Πράγματι λοιπόν πάρα πολλές ε, τροπολογίες, αλλά γιατί είναι και πάρα πολύ σημαντικό το θέμα και επίμαχο σε πολλά κράτη-μέλη. Να το δώρο λοιπόν τι είναι για να μετράμε αν είμαστε 20% αυτό. Το Συμβούλιο, όσο εμείς επεξεργαζόμαστε αυτή την πρόταση, επεξεργάζεται και αυτό διάφορες άλλες ε, λύσεις. Θα ήθελα το Κοινοβούλιο, το έχω ξαναπεί, να δείξει ότι υπάρχει μεγάλη συνένεση μεταξύ μου αλλά και του Συμβουλίου, γιατί τελικά βέβαια τα κράτη-μέλη είναι αυτά τα οποία θα πρέπει να εφαρμόσουν τα μέτρα για τις εξοικονομήσεις, για την ενεργειακή απόδοση. Και εμείς αυτό το οποίο θέλουμε είναι να μειωθεί η χρήση της ενέργειας ώστε αυτό να είναι και προσιτό για εμάς, για τους πολίτες μας, για τις επιχειρήσεις των χωρών μας. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει, να είναι ε, σε προτεραιότητα τα πιο αποδοτικά και τα πιο οικονομικά μέτρα. Και αυτά, σε αυτά τα μέτρα θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στα διάφορα κράτη-μέλη. Χαίρομαι που την προσέγγιση μου την στηρίζουν και άλλοι συνάδελφοι, ιδίω ε, στο άρθρο 10 για τη συμπαραγωγή. Σίγουρα είναι πολύ σημαντική η ενεργειακή απόδοση. Αυτή όμως που θα υποφελούνται από τα μέτρα θα πρέπει να είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν και τις προσπάθειες. Σε ό,τι αφορά τους συμβιβασμούς, νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε πολλά πράγματα υπόψη μας. Ε, το ΕΛΚ είπε πολύ καλά ότι κάποιες συμβιβαστικέ προτάσεις δεν είναι και τόσο συμβιβαστικέ. Δεν προσπαθούν να συμπεριλάβουν όλες τις σχετικές τροπολογίες και υπάρχουν σίγουρα πολύ διαφορετικές απόψεις. Νομίζω ότι θα πρέπει ίσως να ψηφίσουμε όταν υπάρχουν τόσο μεγάλες αποκλήσεις για να δούμε προς τα που κλείνει η πλειοψηφία. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει ευελιξία στα κράτη-μέλη για την εφαρμογή των μέτρων. Εναλλακτικέ λύσεις ό,τι αφορά αυτό το 3% για τα δημόσια κτίρια στην περιφέρειά μου έχω έρθει σε επαφή με το 50% των δημόσιων αρχών για να δω την άποψή τους. Ε, κάποιε μπορούν να τηρήσουν το στόχο του 3%, κάποιε αρχέ το έχουν ήδη κάνει, για άλλε θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αν λοιπόν υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι για την επίτευξη του ίδιου αποτελέσματος στα κράτη-μέλη, αν μπορούν δηλαδή ε, να στοχεύσουν εκεί που θα έχουν το μεγαλύτερο όφελος, να μπορούν να το πράξουν, να υπάρχει ευελιξία. Επίσης, ό,τι αφορά τις τροπολογίες για ε, την αύξηση του χρονοδιαγράμματος. Οι επιχειρήσεις που καταναλώνουν ενέργεια επικεντρώνονται ήδη στα τιμολόγια. Χρειάζονται χρόνο για να μπορέσουν να εφαρμόσουν τα συμπεράσματα των ελέγχων. Πρέπει να δούμε και αυτό το θέμα. Επίσης, ένα άλλο επίμαχο άρθρο είναι το άρθρο 3. Υπάρχουν διαφορές απόψεων. Μιλάμε για εξοικονόμηση, μιλάμε για αποδοτικότητα, μιλάμε για ένταση ενέργειας. Εγώ καταλαβαίνω, καταλαβαίνω απόλυτα το μήνυμα που στέλνουν οι επιχειρήσεις. Αν εμείς ε, αυξανόμαστε και βελτιωνόμαστε, δεν θέλουμε να έχουμε και μεγαλύτερο λογαριασμό να πληρώσουμε, αν έχουμε μεγαλύτερη παραγωγή. Ίσως μπορεί να βρεθεί ένας διαφορετικός συμβιβασμός. Να δούμε δηλαδή το σκέλος της εξοικονόμησης ε, ε, στα κτίρια είτε γραφείων είτε κατοικιών. Τα τρία τέταρτα περίπου της ενέργειας που καταναλώνεται ε, στην ε, Ευρώπη μας έχει δώσει κάποια στοιχεία σχετικά η Κομισιόν. Στο βιομηχανικό τομέα λοιπόν, αν δούμε τώρα το τελευταίο τέταρτο αυτό που έχει να κάνει με τη μεταποίηση, την βιομηχανική παραγωγή, εκεί θα πρέπει να δούμε τη δυνατότητα εξοικονόμηση έντασης, σε ένταση ενέργειας. Ίσως μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα με το άρθρο 3. Να δούμε δηλαδή τα δύο διαφορετικά αυτά μέρη της οικονομίας υπό διαφορετικό πρίσμα. Εσύ ξέρω ότι θέλεις να ισχύσει ο ίδιος κανόνας σε, σε όλο το φάσμα, το 20%. Και ένα άλλο θέμα που με απασχολεί είναι η μελέτη επιπτώσεων. κ. Τσίτσεστερ έκανε πολύ σημαντική δουλειά για το θέμα αυτό των μελετών επιπτώσεων. Νέες ιδέες ε, ω τροποποίηση ενό κειμένου αρχικού της Κομισιόν. Νομίζω ότι εισάγουμε νέε ιδέε. Θα μπορούσαν όμως αυτές να είναι καλές, να πανηρές, να μην έχουν το όφελο που επιδιώκουμε. Εκεί θα πρέπει να γίνουν μελέτε επιπτώσεων. Η Επιτροπή ΙΜΚΟ αυτή τη στιγμή επεξεργάσετε μια πρόταση νομίζω για τις μηχανές και έχουν ε, στείλει μια ανεξάρτητη μελέτη επιπτώσεων. Πρέπει να το κάνουμε και εμείς. Αλλάζουν ε, ίσως ιδέες ή προσεγγίσεις σε κάποια θέματα, αλλά δεν έχουμε κάτι ρηξικέλευθο για να χρειαστεί μια μελέτη επιπτώσεων στο 80% του κειμένου, αλλά μπορεί στο 20% να υπάρχουν ιδέες τέτοιες. Θα έχουμε την 1η Ιανουαρίου το νέο τμήμα ε, του Κοινοβουλίου, νομίζω για τις μέλες επιπτώσεων, θα έχουμε την ομάδα αυτή του Κοινοβουλίου και θα μπορούσαμε να δούμε αυτές τις τροπολογίες, να τους τις διαβιβάσουμε για να δουν αν συνιστούν προσθέμενη αξία. Πάντως πρόοδο σημειώνουμε και θα συνεχίσω και εγώ και όλοι μας φαντάζομαι να εργαζόμαστε σκληρά. Ευχαριστώ. Κυρία Χολ, ευχαριστώ πολύ. Ξεκινώ με κάποια σημεία σε απάντηση σε αυτά που είπε και η Βίκη μόλις τώρα για την αξιολόγηση επιπτώσεων. Νομίζω ότι πρέπει καταρχήν να αποφασίσουμε ε, τι θα γίνει με το κείμενο στην Επιτροπή ε, Ήτρε και θα επανέλθω σε αυτό σε λίγο. προσπαθώντας να δούμε τι κάνει το Συμβούλιο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εμείς είμαστε Κοινοβούλιο και εκείνη είναι Συμβούλιο και αυτός είναι και ο σκοπός των τριμερών διαλόγων. Νομίζω αργότερα θα πρέπει να ασχοληθούμε με το τι κάνει το Συμβούλιο. Απογοητεύτηκα κάπως από τα σχόλια που έγιναν για τη δουλειά των σκιωδών και το χρονοδιάγραμμα. Νομίζω ότι είναι πολύ συστηματική η δουλειά και έχει προγραμματιστεί πάρα πολύ καλά και αν συνεχίσουμε κατά αυτόν τον τρόπο θα τα καταφέρουμε μια χαρά με το χρονοδιάγραμμα. Και πιστεύω ότι είναι σημαντικό να μην υπάρχει καμία αμφιβολία για τους συναδέλφους, γιατί αυτό δεν βοηθάει τον προγραμματισμό μας. Το γεγονός ότι είμαστε σήμερα λίγο πριν από τα Χριστούγεννα αποδεικνύει ότι παίρνουμε πολύ στα σοβαρά τη δουλειά μας, όπως και θα έπρεπε εξάλλου. Το ότι δεν θέλουμε να δουλεύουμε με πολλές τροπολογίες είναι κάτι το οποίο δεν είναι δίκαιο να το λέμε. Οι σκιώδεις συγητές ευχαρίστως θέλουν να δουλέψουν για να καταλήξουμε σε καλά συμβιβαστικά κείμενα. Αυτό που ανέφερε η κυρία Φόρντ είναι σωστό. Αν δεν υπάρχει πολιτική συμφωνία θα πρέπει ξεκάθαρα να το πούμε. Να μην προσποιούμεθα ότι κατά κάποιο τρόπο οφείλεται η αποτυχία στο ότι δεν αφιερώσαμε χρόνο για συμβιβαστικέ τροπολογίε κάθε άλλο. Νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε αυτό που κάναμε, γιατί δουλεύουμε σοβαρά και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε σοβαρά και να αφιερώνουμε το χρόνο ο οποίος απαιτείται. Και σίγουρα και ο Πρόεδρος θα συμφωνεί. Ας δούμε γιατί υπάρχει αυτή η οδηγία, γιατί χανόμαστε στις λεπτομέρειες και ξεχνάμε το γιατί υπάρχει αυτή η οδηγία. Ο πιο σημαντικός λόγος για την οδηγία αυτή είναι ότι παραμένει ο στόχος της αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος όπως αποφάσισαν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων το 2007 και θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή. Αν κάποιος πιστεύει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα κλιματικής αλλαγή, ας το πούμε καλύτερα παρά να μπαίνουμε σε λεπτομέρειες τη οδηγία και να λέμε ότι αυτά μας φταίνε. Μα ανησυχεί η κλιματική αλλαγή, αλλά αυτή τη στιγμή μα ανησυχεί πάρα πολύ η οικονομική κατάσταση στην Ευρώπη. Και αυτή η οδηγία θέλουμε να αυξήσει το ΑΕΠ και επίσης ε, με αυτή την οδηγία 200 δις λιγότερα θα δαπανώνται για την ενέργεια κάθε χρόνο. Πράγμα το οποίο σίγουρα θα βοηθήσει την οικονομία. Δεν συμφωνώ με τα σχόλια που έγιναν προηγουμένως ότι θα μπορούσαμε να το κάνουμε καλύτερα εάν υπήρχε ε, ένας στόχος ε, για την ένταση ε, της βιομηχανίας περισσότερο παρά για την εξοικονόμηση ενέργειας. είναι πιο δύσκολο για τις επιχειρήσεις ε, να εκπληρώσουν ένα στόχο έντασης ενέργειας από ότι εξοικονόμησης ενέργειας. Δεν θα βοηθούσαμε λοιπόν τις εταιρείες μας αν θέταμε ένα τέτοιο στόχο. Θέλουμε να επιτύχουμε την εξοικονόμηση του 20% το 2020 και νομίζω ότι αν θέσουμε το στόχο της έντασης ενέργειας δεν θα τα καταφέρουμε. Όσον αφορά την ευελιξία, Πιστεύω ότι είναι σημαντική η ευελιξία και υπάρχουν αρκετά άρθρα όπου μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση γιατί και στα 27 κράτη-μέλη η πολιτική που ακολουθείται είναι διαφορετική. Κάνουμε τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο. Είναι δύσκολο να βρούμε ένα κείμενο και δεν τα καταφέρνει και η Επιτροπή να βρει ένα κείμενο που θα καλύπτει όλες τις διαφορετικές περιστάσεις των κρατών μελών. Και όταν μιλάμε για το 1,5% ετησίως, είναι σημαντικό να δούμε ότι υπάρχουν άρθρα που προτείνουν ένα διαφορετικό τρόπο για να το επιτύχουμε. Και το 3% ε, επιφάνειας ε, ετησίως για την ανακαίνιση δημοσίων χώρων δεν νομίζω ότι και αυτό είναι το σημαντικότερο. Πρέπει να δούμε ε, αν οι δημόσιες αρχές μειώνουν την ενέργεια ετησίως καταβάλλοντας προσπάθειες χωρίς να πούμε ότι θα είναι 3% της επιφάνειας υποχρεωτικά. Υπάρχει η δυνατότητα να δώσουμε μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη-μέλη εφόσον έχουν συμφωνήσει τα κράτη-μέλη με τους δεσμευτικούς στόχους. Συμφωνώ με τους συναδέλφους ότι δεν πρέπει να κολλάμε στις λεπτομέρειες, αλλά να μην ξεχνάμε και τους στόχους της οδηγίας. Συνδυασμός λοιπόν δεσμευτικών στόχων και ευελιξίας πιστεύω ότι είναι η σωστή πορεία. Σχετικά με τις δημόσιες ε, συμβάσεις, ε, εδώ είναι κάπως περίεργα τα πράγματα, γιατί νομίζω ότι σήμερα περιμένουμε από την οδηγία την έκδοση της οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις. Να προσέξουμε λοιπόν πάρα πολύ αυτά τα οποία κάνουμε εδώ για τις δημόσιες συμβάσεις να ταιριάζουν με την οδηγία που ετοιμάζει τώρα η Επιτροπή. Και να μην ξεχνάμε γιατί είναι σημαντικός ο τομέας των δημόσιων συμβάσεων. Διότι ε, κινητοποιεί την αγορά για την εξοικονόμηση ενέργειας, μειώνει τις τιμές και κάνει εξοικονόμηση δημοσίου χρήματος μακροπρόθεσμα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο σίγουρα θα είναι στόχος και της οδηγίας για τις δημόσιες προμήθειες. Τέλος, σχετικά με τον οδικό χάρτη για το 2050 και το 80% των κτηρίων ε, που θα πρέπει να έχουν ενεργειακή αποδοτικότητα μέχρι το 2050. Μπορεί να έχουμε πεθάνει μέχρι τότε βέβαια. δεν θα πρέπει να σκεφτόμαστε αυτό, αλλά να σκεφτόμαστε ότι αυτό που κάνουμε σήμερα είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να επηρεάσουμε το αύριο. Έχουμε τεράστια ε, προσπάθεια για να μην έχουμε εκπομπές διοκτήτου του άνθρακος μέχρι το 2050, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει τώρα να καταβάλουμε πολλά βήματα και μπορεί να μην ζούμε εμείς το 2050, θα ζουν όμως τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας και θα ήθελα να ζουν ε, με σωστό τρόπο και να μην έχουμε συμβάλει εμείς με τη σπατάλη ενέργειας σε αρνητική διαμόρφωση του μέλλοντος. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βιντάλ Κουάντρας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αφού άκουσα όλες τις παρεμβάσεις, νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι ήρθε το πληρώνο του χρόνου να έχουμε μια ρεαλιστική προσέγγιση στη συζήτηση αυτή. Γιατί Όλοι ξέρουμε ότι το να έχουμε ένα καθολικό δεσμευτικό στόχο είναι κοκκίνη γραμμή για το Συμβούλιο. Επομένως, φαίνεται ότι είναι πιο παραγωγικό να επικεντρωθούμε στα μέτρα. Και να προσπαθήσουμε να εκπονήσουμε όσο το δυνατό καλύτερα μέτρα, επιτρέποντας φυσικά και την απαραίτητη ευελιξία για τα κράτη-μέλη για να αποδείξουν μέσω των εθνικών σχεδίων τους ότι και άλλα μέτρα θα είναι ισοδύναμα για την επίτευξη των εθνικών στόχων. Τώρα, για να περάσω σε πιο συγκεκριμένα σχόλια σε σχέση με το άρθρο 3, θέλω να προτείνω μια συμβιβαστική οδό. Ίσως αν διατηρήσουμε το άρθρο όπως είναι αυτή τη στιγμή, όπως το προτείνει η Κομισιόν, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε ένα τμήμα που να λέει ότι όταν ε, μιλάμε για τους ενεργοβόρους τομείς, εντατικούς τομείς ενέργειας, θα πρέπει τα κράτη-μέλη να έχουν ένα στόχο ε, σε σχέση με την εντατικότητα της ενέργειας, ε, σε σχέση με το ΕΠ, όπως πρότεινε η κυρία Φόρντ. Νομίζω ότι αυτό είναι καλός τρόπος να πετύχουμε συμβασμό. Έτσι θα διατηρήσουμε τους εθνικούς στόχους, έτσι όπως εκφράζονται με όρους απόλυτης μείωσης της κατανάλωσης και αποφεύγουμε και τη ζημία των τομέων αυτών που είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στο θέμα της ε, τιμής της ενέργειας. Σε σχέση με το άρθρο 6, θέλω να κάνω δύο σύντομα σχόλια. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στην ευελιξία στο άρθρο αυτό. Δηλαδή, να πούμε ότι η δυνατότητα για ένα κράτος μέλος να αποδείξει ότι και άλλα μέτρα που συμπεριλαμβάνονται στο σχέδιό του είναι ισοδύναμα για να πετύχει τους στόχους της ενεργειακής αποδοτικότητας χρησιμοποιώντας το άρθρο 69. Δεν καταλαβαίνω γιατί κάτι τέτοιο θα πρέπει να υπόκειται σε μία και μόνο υποχρέωση υποβολή έκθεση των Κομισιόν, όπω λέγεται τώρα στο άρθρο. Δεν θα πρέπει να έχουμε διπλές υποχρεώσει υποβολή ε, εκθέσεων. Έτσι λοιπόν θα πρότεινα οποιοδήποτε άλλο μέτρο να υπόκειται στο άρθρο 6 και στη σχετική υποχρέωση υποβολή εκθέσεων ε, όταν τα κράτη-μέλη υποβάλλουν όλα τα εθνικά του σχέδια ενεργειακή αποδοτικότητα στην Κομισιόν. Και αυτό να αρκεί. Και να μην έχουμε επικάλυψη αυτών των υποχρεώσεων. Πολλοί βουλευτές καταθέσαμε μέτρα που διευκολύνουν την ενεργή συμμετοχή των καταναλωτών ε, στην ε, ενεργειακή αποδοτικότητα. Για να επιτρέψουμε κάτι τέτοιο θα πρότεινα το άρθρο 6 παράγραφος 3 να αναφέρει το εξής. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εκφράζουν ε, το ποσό της χρησιμοποιημένης ενέργεια που απαιτείται από κάθε μέρος με όρους τελικής ενέργειας ή και, πρωτογενούς, ή και κατανάλωσης πρωτομεριανούς ενέργειας. Αυτή η συμπερίληψη, καταναλωσης ενεργειας αυτη αυτή η ε, διατύπωση είναι πιο καθολική και δίνει στα κρατημέλη και τη δυνατότητα να θέσουν προτεραιότητα είτε τελική εξοικονόμηση ενέργειας είτε στην πρωτογενή ενέργεια. Κατόπιν να είμαι ικανοποιημένο ε, με τη διατύπωση πιθανών συμβιβασμών ε, στο σημείο 10 που εξετάζουμε τώρα. Αλλά θέλω και εδώ να κάνω δύο σύντομα σχόλια. Σε ορισμένε ε, παραγράφους εξακολουθεί να αναφέρεται η τηλεθέρμανση και η τηλεψήξη. Και θέλω να υπενθυμίσω στον εισηγητή, στον κύριο Τούρμες και στους υπόλοιπους κοιόδης, ότι η τηλεθέρμανση και η τηλεψήξη είναι μια περιορισμένη έννοια. Γιατί η CHP, η συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας, είναι κάτι ευρύτερο από την τηλεθέρμανση και την τηλεψήξη. Έτσι λοιπόν θα έπρεπε να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση. Θα μπορούσαμε να λέμε λοιπόν συμπαραγωγή ή απλώς θέρμανση και ψήξη, όχι τηλεθέρμανση και τηλεψήξη. Και με αυτόν τον τρόπο συμπεριλαμβάνουμε όλα τα είδη της συμπαραγωγής και όχι μόνο την τηλεθέρμανση και την τηλεψήξη. Αυτό είναι κάτι που εγώ θεωρώ ουσιαστικό. Δεύτερον, Ξέρω ότι πρότεινε ο εισηγητης είναι ένα νέο παράρτημα 8α για να καθοδηγήσει την Κομισιόν από το 2013 και μετά σε της πράξη να εκπονήσει τους όρους ε, ε, για το να υπάρχει μία ανάλυση κόστους ωφέλους. Εγώ υποστηρίζω κάτι τέτοιο για οποιοδήποτε μέτρο στην παραγωγή ληφθεί, αλλά έχω μια αμφιβολία ότι η οδηγία είναι το κατάλληλο σημείο για να προσδιορίσουμε το περιεχόμενο μιας τέτοιας ανάλυσης κόστους ωφέλους. Νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε και να δούμε τι θα μας παρουσιάσει η Κομισιόν μέσω της κατεξουσιοδότης πράξης. Σε ό,τι αφορά τα άρθρα 4 και 5, έχω ένα σημείο που θέλω να καλωσορίσω στις συζητήσεις αυτές το γεγονός ότι πέρα από τις ανακαινήσεις των κτηρίων, τα κράτη-μέλη μπορούν να λάβουν και εναλλακτικά μέτρα για να μειώσουν 3% ετησίως την ενεργειακή κατανάλωση. Φυσικά, ορισμένοι από εμά θα μπορούσαν να συζητήσουν το αν το 3% είναι υπερβολικό ή όχι, αλλά η αρχή θα πρέπει να είναι ευπρόσδεκτη. Γιατί υπάρχει κάποια σύγχυση στο ότι η ενεργειακή απόδοση ενός κτηρίου μπορεί να βελτιωθεί μόνο μέσω της ανακαίνησης. Αλλά υπάρχουν ε, και άλλες ε, πιθανές συσκευές ή υπηρεσίες ενεργειακής αποδοτικότητας που θα μπορούσαν να βελτιώσουν την αποδοτικότητα χωρίς ε, να χρειάζεται μεγάλη ανακαίνιση. Και τέλος, ένα πολύ σύντομο σχόλιο για το αφροκτό για τους εξύπνους μετρητές. Πιστεύω ότι θα πρέπει να σκεφτούμε περισσότερο το πιθανό κόστος των μέτρων αυτών. Έτσι λοιπόν, εγώ θα ήθελα να σας καλέσω να συμπεριληφθεί η τροπολογία μου που καλεί υποχρέωση για φύσεις μετρητές όπου είναι τεχνικά ε, δυνατό και αποτελεσματικός προς το κόστος για τον επενδυτή. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι βρισκόμαστε σε πάρα πολύ επικοδομητικές συζητήσει και νομίζω ότι το αποτέλεσμα θα είναι καρποφόρο. Ευχαριστώ. Κύριε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχω ανάμεικτα συναισθήματα με βάση τη συζήτηση αυτή. Νομίζω ότι κάποιοι συνάδελφοι ορισμένες φορές δεν ξέρουν ακριβώς γιατί μιλάνε. Αν δει κανεί ε, τους δεσμευτικούς στόχους, εδώ μιλάμε για 20%, όχι όμως για μείωση 20% στη χρήση ή 20% αύξηση στην απόδοση. Και τι θα πει απόδοση, πώς μετράτε η απόδοση, πώς ποσοτικοποιείται σίγουρα πρέπει να ποσοτικοποιηθεί διαφορετικά στους τομείς της κατασκευής, ε, της βιομηχανίας, χαλιβουργία ε, κτλ. Κατά περίπτωση δηλαδή να υπολογίζεται με επιστημονικά κριτήρια και με ένα συγκεκριμένο ποσοστό. Αναχώρα όμως πολιτικός στόχος για τις ε, κυβερνήσεις 20% αύξηση στην ενεργειακή απόδοση. Αυτό θα πρέπει να υπολογιστεί ως διαφορά μεταξύ της χρήσης, όπως τη μετράει η Eurostat, διά του ΑΕΠΑ. ...99-2020, αυτά τα χρόνια. Δηλαδή να διαιρείται με το ΑΕΠ της ε, χρονιάς εισόδου και να ισχύει μετά το ποσοστό. Εκεί μπορούμε να δούμε την αποδοτικότητα. Έχω λοιπόν να κάνω την εξής πρόταση στον κύριο Τούρμες. Δεν μπορώ να πω ότι συμφωνώ με τις τροπολογίες σας, κύριε Τούρμες, εκεί που λέτε ότι η αύξηση στην απόδοση ισούται ουσιαστικά με τη μείωση στη χρήση. Συμφωνώ με τον κύριο Πίπερ, που λέει ότι δεν μπορούμε να μειώσουμε την χρήση αν δεν επενδύσουμε στην αύξηση της απόδοσης. Αλλά είναι δύο διαφορετικά πράγματα αυτά. Μπορείτε κύριε Τούρβες να φανταστείτε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αυξάνει την ενεργειακή απόδοση περισσότερο από το 20% από τώρα μέχρι το 2020 ενώ ταυτόχρονα αυξάνει και τη χρήση της ενέργειας. Διότι έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες άλλες περισσότερο και άλλες λιγότερο αναπτυγμένες που πρέπει να αναπτυχθούν. Και όλα αυτά βέβαια συνεπάγονται χρήση ενέργειας. αλλά και ενεργειακή απόδοση μπορεί να αυξηθεί. Μπορούμε να μετρήσουμε την ενεργειακή απόδοση με πολλούς τρόπους, αλλά τον, ε, ορισμό αυτό ε, νομίζω ότι πρέπει να τον επεξεργαστούμε πολύ σωστά για να αποφύγουμε παρανοήσεις. Η κυρία Μέρκης τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Λίγα θέματα θέλω να αναφέρω στο πλαίσιο της οδηγίας αυτής, πρώτα απ' όλα πεδίο εφαρμογή. Αλλά αυτό ήδη πολλές φορές το έχουμε συζητήσει. Όπως όμως και πολλοί συνάδελφοι, έτσι και εγώ έχω την εντύπωση ότι πρέπει να επεκτείνουμε το πεδίο εφαρμογή και να μην καλύπτονται μόνο τα δημόσια κτίρια, αλλά και άλλοι τομείς. Και ιδίω να λαμβάνουμε υπόψη και τους ενοικιαστές, τους πλέον ευάλωτους ενοικιαστές, οι οποίοι θέλουν να είναι ζεστό το σπίτι τους το χειμώνα. Αν επεκτείνουμε το πεδίο εφαρμογή βοηθώντας τα άτομα αυτά, νομίζω ότι θα ωφελήσουμε και την οικονομία γιατί θα προωθήσουμε τις επενδύσεις και θα βοηθήσουμε την επίτευξη στόχων που δεν είναι δεσμευτικοί, αλλά θα πρέπει να γίνουν δεσμευτικοί. Πάντως νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μια επιλογή, είτε το ένα είτε το άλλο. Αν τα κράτη-μέλη δεν θέλουν να στηρίξουν τους δεσμευτικούς στόχους, φυσικά θα πρέπει να δώσουμε περισσότερες εμείς υπαγορεύσεις και κατευθύνσεις. Αλλά καλό θα ήταν να, υπάρχουν, να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία σε ό,τι αφορά την υλοποίηση των μέτρων περί ενεργειακής απόδοσης. Γιατί κάθε κράτος μέλος είναι διαφορετικό και δεν θα πρέπει να είμαστε υπερβολικά λεπτολόγοι, λεπτομεριακοί για τα κράτη-μέλη σχετικά με το πώς θα πρέπει να εφαρμόσουν αυτά τα μέτρα. Ναι, μεν δεσμευτική στόχη, ναι, ενεργειακή απόδοση στο μέγιστο δυνατό βαθμό, αφήνοντας όμως περιθώρια για τα κράτη-μέλη. Αφήνοντας κάποιο ελεύθερο χώρο για να κινηθούν. Και ένα πάρα πολύ σημαντικό για μένα θέμα πάρα πολύ συχνά εστιάζουμε στις μεγάλες λύσεις, αλλά σας παρακαλώ να προσέξουμε και τις μικρές λύσεις. Ενεργειακή απόδοση μέσω, παραδείγματο χάρη, ε, της ε, μικροπαραγωγής, της μικροσυμπαραγωγής σε τοπικό επίπεδο. Ο Επίτροπος Αρμόδης για την Ενέργεια δεν νομίζω ότι προσέχει και πολύ το γεγονός ότι ο αριθμός ε, πολλών μικρών μονάδων μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο. Ε, να φτιάξει ένα μεγάλο σύνολο. Επίσης θα πρέπει να ανταποκριθούμε στη ζήτηση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μέχρι στιγμή η αγορά ενέργειας δεν μπορεί να καλύψει. Θα πρέπει λοιπόν να τροποποιήσουμε την υποδοχή και την υποδομή συγγνώμη, και την αγορά ενέργειας κατά τρόπο ώστε να υπάρχει μέγιστη δυνατή ευελιξία για τους ε, πελάτες. Και ένα τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό θέμα. Θα το ξανασυζητήσουμε με τον κύριο Τούρμες αυτό. Θα ήθελα οι καταναλωτές οι οποίοι ανατροφοδοτούν το δίκτυο να τους επιστρέφεται η τιμή λιανικής. Θα το συζητήσουμε βέβαια. Απλά θα ήθελα να μου απαντήσει ο κύριος Τούρμες όλα αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Επιτρέψτε μου να προσθέσω κάτι σε σχέση με αυτά που είπε και η κυρία Μέρκης, για να τα σκεφτούμε απλώ. Εγώ δεν είμαι υπέρ των δεσμευτικών στόχων κλπ. Αλλά, εν περιπτώσει, όσο ακούω αυτά που λέγονται, σκέφτομαι μήπως είναι σκόπιμο να έχουμε ένα δεσμευτικό στόχο και για τα συγκεκριμένα μέτρα να αφήσουμε τα κράτη-μέλη να αποφασίσουν τι θέλουν να κάνουν. Αυτό το, επιχείρημα που ακούω ε, και το άκουσα και από τον Επίτροπο τον κύριο Έτινγκ είναι ότι τα κράτη-μέλη δεν θα συμφωνήσουν. Αποφασίζουμε εμείς ως Κοινοβούλιο το τι θα αποφασίσει το Συμβούλιο ή αποφασίζουμε εμείς τι θέλουμε εμείς ως Κοινοβούλιο. Γιατί πάντοτε ε, γίνεται μια συζήτηση επειδή το Συμβούλιο έχει κάποια συγκεκριμένη άποψη. Εμείς τη δική μας θέση πρέπει να υπερασπιστούμε. Συγγνώμη, αλλά ήθελα να το κάνω αυτό το σχόλιο. Κύριο Σκέλη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Τούρμες και ευχαριστώ και όλους ε, για την ε, συνεισφορά του σήμερα το πρωί. Αν έχουμε στόχους για το 2020 και για το 2050, θα πρέπει να τους επιτύχουμε. Το πώς θα τους επιτύχουμε είναι ένα θέμα που θα το επεξεργαστούμε τις κατάλληλες λεπτομέρειες. Θα πρέπει να κάνουμε μια αξιολόγηση κάθε δύο-τρία χρόνια για να δούμε πώς πορευόμαστε και να κάνουμε τις απαραίτητες προσαρμογές, γιατί αν δεν επιτύχουμε αυτούς τους στόχους υπονομεύουμε όλες τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ήδη με την στρατηγική της Λισαβόνας ε, είδαμε ότι δεν ήταν ικανοποιητικά αυτά που επιτύχαμε. Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για μεγαλύτερη αποδοτικότητα της ενέργειας και εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση της οικονομίας. Όταν θα έχουμε ανάκαμψη της οικονομίας, σίγουρα θα υπάρξει αυξημένη ζήτηση ενέργειας και θα πρέπει και αυτό να το λάβουμε υπόψη μας. Ταυτόχρονα, εάν έχουμε συγκεκριμένους στόχους, θα πρέπει να υποχρεωθούν όλοι ε, να φροντίσουν να τους επιτύχουν αυτούς τους στόχους. Αυτό θα δημιουργήσει και καλύτερη αγορά και θα δώσει μεγαλύτερη σημασία στην έρευνα για να έχουμε πιο, πιο αποδοτικά αυτοκίνητα παραδείγματος χάρη. θα πιέσουμε και τη βιομηχανία να συμμορφωθεί με τα πρότυπα αποδοτικότητας που θα έχουμε θέσει εμείς με συγκεκριμένα χρονοδιογράμματα. Το ίδιο ισχύει και για τα κτίρια. Και στη δική μου εκλογική περιφέρεια έχω πολλούς κατασκευαστές κτίριων που έχουν ε, πιστοποιημένα κτίρια με ενεργητική αποδοτικότητα και έχουν ε, και συμβάσεις στη Μέση Ανατολή γιατί ε, φαίνεται ότι η τακτική τους για την πιστοποίηση ενεργητικά αποδοτικών κτηρίων είναι αποδοτική. Δεν θα πρέπει να επιτρέπουμε την κατασκευή κτηρίων που δεν είναι ενεργειακά αποδοτικά και για τα δημόσια κτίρια, ιδίως τα κτίρια που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση, ε, θα πρέπει να τηρούνται αυτές οι αρχές το μήνυμα της κλιματικής αλλαγής και το μήνυμα της ενεργειακής αποδοτικότητας είναι ένα μήνυμα που σιγά σιγά αρχίζει να γίνεται κατανοητό και αποδεκτό από την κοινή γνώμη. Και ιδίω, όπως είπε ο κύριο Τούρμες, αν μπορεί να είναι ευθυνότερο ο ηλεκτρισμό, τόσο το καλύτερο. Θα πρέπει να επιτύχουμε τους στόχους μας και για περιβαλλοντικούς σκοπούς και για καθαρά πρακτικούς σκοπούς και ανάπτυξη της οικονομίας της Ευρώπης. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Καβάλιο. Ε, Ευχαριστώ. Θα επικεντρωθώ στο άρθρο 3. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να δούμε και τους στόχους ε, κατανάλωσης αλλά και το στόχο έντασης ενέργειας, ε, πώς ε, θα γίνει η κατανομή σε κάθε κράτος μέλος. Και ανησυχώ κυρίως για κράτη-μέλη, στον οποίο το ΕΠ θα μειωθεί. Και έχουμε και πρόβλεψη ότι στο δικό μου κράτος μέλος θα έχουμε μείωση του ΕΠ. Το επόμενο τουλάχιστον ένα-δύο έτη. Και έτσι λοιπόν πρέπει να ξέρουμε εδώ πώς ακριβώς θα εξελιχθεί αυτό το θέμα και τις συνάγκες των κρατών μελών μας και πώς τις μεταφράζουμε. Το δεύτερο σχόλιο. Νομίζω ότι η πρόταση της κυρίας Φόρτ ήταν παρομοία με αυτό που πρότεινε ο κύριος Ζιδαλκουάδρα. Να έχουμε δηλαδή ένα στόχο κατανάλωσης για την οικονομία γενικά πέρα από τη βιομηχανία και έχουμε και ένα στόχο έντασης για τη βιομηχανία. Νομίζω ότι η κυρία Φορτ μίλησε γενικά για τη βιομηχανία και ο Βιδάλ Κουάδρας ε, ε, μίλησε για την ε, ενεργοβόρο βιομηχανία. Θα πρέπει να το δούμε αυτό αλλά θα μπορούσαμε να έχουμε ένα συμβασμό και ως στόχους κατανάλωσης για τα κτίρια και για όλους τους τομείς πέραν της βιομηχανίας. Θα πρέπει ε, να καταναμηθούν χώρες, και επίσης ε, ο στόχος έντες ενέργειας θα πρέπει να εξεταστεί ένα τομέα. Και θα πρέπει να έχουμε ένα μοντέλο, να προκύψουν κάποια αποτελέσματα από αυτό, να εξετάσουμε τα αποτελέσματα και να δούμε ποια είναι τα αριθμητικά στοιχεία και πώς έχει η κατάσταση γιατί αποφασίζουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό για το μέλλον της οικονομίας μας. Έχω μια ερώτηση λοιπόν, αν τα δύο άτομα που το πρότειναν αυτό ή η Κομισιόν, αν ε, μπορούν να μας δώσουν κάποια αριθμητικά στοιχεία, δηλαδή πώς θα μοιάζει η λύση αυτή, πώς θα διαμορφωθεί, γιατί θα μπορούσε να αποτελέσει μια συμβαστική λύση για την επιλύση αυτού του προβλήματος. Είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο, αλλά είναι πολύπλοκη και η πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν μάλλον και η λύση δεν μπορεί να είναι απλή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις νομίζω ότι εδώ έχουν μια μεγάλη ευκαιρία εάν ε, μπορούμε να θέσουμε συγκεκριμένους στόχους σε συγκεκριμένους τομείς. Και θα πρέπει να προετοιμαστούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις για πολλές δραστηριότητες ε, που θα χρειαστούν και για την κατάλληλη κατάρτιση που θα χρειαστούν για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα. Και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας μπορεί να παράσχει εδώ ε, βοήθεια. Γιατί ε, εδώ νομίζω ότι είναι πολλά τα θετικά σημεία και στο άρθρο 3 θέτει δεσμευτικούς στόχους, πράγμα το οποίο είναι θετικό. Δεν θα πρέπει όμως να υπάρχει η απειλή κυρώσεων. Θα πρέπει να υπάρχουν δεσμευτικοί στόχοι και τα κράτη-μέλη να ακολουθούν συστήματα βέλτιστων πρακτικών και συγκρίσεων benchmarking, ούτως ώστε να επιτύχουν αυτό το οποίο είναι κατά το καλύτερο δυνατό τρόπο εφικτό έχουμε το στόχο για το 2020 και πρέπει να δούμε πώς μπορούμε, αυτός ο στόχος ε, ε, μπορεί να, με τους, ε, να συνδυαστεί με τους στόχους των μεταγενέστερων ετών. Στο άρθρο 6 για την ενεργειακή αποδοτικότητα θέλω να πω ότι το παράρτημα 5 περιλαμβάνει πολλά γραφειοκρατικά στοιχεία και θα πρέπει ο κύριος Στόιμπε με την ομάδα του να προσπαθήσει να εξετάσει αν όντως ε, είναι απαραίτητα όλα αυτά και θα πρέπει και το Κοινοβούλιο να διεξαγάγει την αξιολόγηση επιπτώσεων διότι μας ενδιαφέρει ε, να δούμε ε, κατά πόσο είναι προσαρμοσμένοι οι στόχοι μας και οι ορισμοί με την ε, πραγματικότητα. Ε, γιατί πώς θα το αντιμετωπίσει μια κρατική αρχή αν μια ηλεκτρική συσκευή δεν, είναι, δεν πληρεί τους στόχους που έχουμε θέσει και που ορίζονται βάσει των ορισμών και του παρατήματος. Ε, το πρόγραμμα για την ευθύη ενέργεια θα μπορούσε να είναι μια καλή προσέγγιση και νομίζω ότι εδώ θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει συμπληρωματικές προτάσεις. Η συζήτηση για τα πιστοποιητικά πιστεύω ότι δεν είναι χρήσιμη αυτή τη στιγμή της οικονομικής κρίσης. Δεν θέλουμε να διώξουμε από την Ευρώπη τη βιομηχανία μας που ήδη αντιμετωπίζει δυσκολίες στην Ευρώπη. Μας ενδιαφέρει να βοηθήσουμε μέσω της έρευνας και της καινοτομίας τον τομέα των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακος χωρίς να επιβάλλουμε πρόσθετες επιβαρύνσεις που θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη ανεργία. Αυτό δεν μπορεί να είναι ο στόχος μας αυτή τη στιγμή. θα πρέπει να επιβραβεύσουμε τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται και δεν θα πρέπει ε, να τιμωρείται αυτός ο οποίος έχει αναλάβει δράση σε προημότερο στάδιο. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, στις 11.30 περιμένουμε την Πολωνική Προεδρία βάσει του προγράμματος και έχω άλλες, ε, άλλα έξι ονόματα και έχουμε και την Επιτροπή. Γι' αυτό σας παρακαλώ όλους να είστε σύντομοι για να μπορέσουμε να προλάβουμε. Κυρία Ποδηματά. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ένα γενικό εισαγωγικό σχόλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις παρεμβάσεις των συναδέλφων. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι η ενεργειακή αποδοτικότητα είναι κάτι πολύ σημαντικό και τα ωφέλη που μπορούν να προκύψουν ε, για την πραγματική οικονομία και ιδίω για τις μικρές και μικρές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, δηλαδή από όλους αυτούς ε, που θίγονται από τη σημερινή κρίση. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι στους στόχους μας, τώρα περισσότερο από ποτέ, γιατί πρέπει να προωθήσουμε την ανάπτυξη εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι εκτός Ευρώπης στη Μεσσυνατολή, όπω είπε και ο κύριο Ρούμπιχ πριν. Και φυσικά όλοι αναγνωρίζουμε ότι είναι δύσκολο να βελτιώσουμε την ενεργειακή αποδοτικότητα γιατί χρειάζεται μία επένδυση εκ των προτέρων και τα ωφέλη, αν και είναι εγγυημένα, θα γίνουν αισθητά μετά από αρκετό χρονικό διάστημα. Γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι η χρηματοδότηση είναι πολύ σημαντικό θέμα για την επιτυχία αυτής της οδηγίας. Ε, το ίδιο ισχύει και για την οδηγία νεοσύμων πηγών ενέργειας. Θεωρώ ότι αποτελεί επιτυχία κυρίως ε, λόγω των ε, ε, τιμών fit-in που συμπεριλαμβάνονται εκεί. Τώρα αντιμετωπίζουμε ένα σημαντικό κίνδυνο ε, πιστοτικών ε, επεισοδίων. Διστάζουν οι τράπεζες να δανείσουν τα νοικοκυριά για την πραγματική οικονομία και νομίζω δύο τι να μπορούμε να κάνουμε. Καταρχήν, πιστεύω ότι θα πρέπει να ασκήσουμε κάποια πίεση στην έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να προσδιορίσουν τουλάχιστον κάποιες ξεκάθαρες κατευθυντηρίες γραμμές για το πώς οι ευρωπαϊκές τράπεζες που θα υποφεληθούν από, την τριετή, από το πρόγραμμα χρηματοδότησης με πάρα πολύ χαμηλά επιτόκια, πώς θα δαπανίσουν αυτά τα χρήματα ή τουλάχιστον να διασφαλίσουμε ότι ένα τμήμα αυτών των χρημάτων θα μεταφερθεί με τη μορφή ρευστότητα στην πραγματική οικονομία. Το δεύτερο που μπορούμε να κάνουμε συμπεριλαμβάνεται σε αυτό το σχέδιο πρότασης. Πρόκειται για το νέο άρθρο 2α το οποίο έχει να κάνει με τη δημιουργία νέων χρηματοδοτικών μηχανισμών ε, για την ενεργειακή αποδοτικότητα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι όλες οι φιλόδοξες πολιτικές που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το σχέδιο οδηγία ε, θα υλοποιηθούν. Αν δεν διασφαλίσουμε ότι η χρηματοδότηση της ενεργειακής αποδοτικότητας υπάρχει, δεν θα πετύχουμε τους ε, στόχους για το 2020 ή τουλάχιστον δεν θα τους πετύχουμε με ένα συνεκτικό και συνεπή τρόπο. Και φοβάμαι ότι οι υποχρεώσεις ε, εξοικονόμησης ενέργειας του 1,5% δεν θα αρκέσουν από μόνες της. Και κάτι ακόμα, Πρόεδρε, τελευταίο σημείο, σχετίζεται με τους ευπαθείς καταναλωτές. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα λάβουν στήριξη και υπό τη μορφή προτεραιότητες. Ε, δηλαδή όχι μόνο να επιβολούνται από χαμηλότερους λογαριασμούς ενέργειας στο μέλλον, αλλά να διασφαλίσουμε και ότι δεν θα σηκώσουν το κόστος της ενεργειακής ποδοτικότητας χωρίς να αποφεληθούν ποτέ. Αυτό το τμήμα του πληθυσμού θα βρίσκεται στην πιο δύσκολη θέση να επενδύσει, να συγκεντρώσει χρήματα για επενδύσεις, αλλά έχει πολύ μεγάλο δυναμικό για να συνεισφέρει στο να πετύχουμε την ενεργειακή αποδοτικότητα. Ευχαριστώ. Äh, um Σύντομα παρακαλώ, γιατί μόνο δύο άτομα θα μπορούν να λάβουν το λόγο. Κύριος Μετζάρος. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι τόσο απλό να πούμε κάτι από αυτού, γιατί είναι ένα σύστημα πάρα πολύ πολύπλοκο. Άκουσα με μεγάλο σεβασμό όλες τις παρεμβάσεις. Έπρεπε να είμαι και σε μια ψηφοφορία στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Είναι προτάσεις που θα πρέπει να διαμορφώσουν το μέλλον και να συνεισφέρουμε στην ενεργειακή αποδοτικότητα και να συνδιαμορφώσουν ε, το μέλλον μας. Χαίρομαι λοιπόν που θα έχουμε τη δυνατότητα να συνεργαστούμε για αυτό το θέμα. Και η μελλοντική ε, Δανέζικη Προεδρία έχει εντάξει αυτό το θέμα στις δραστηριότητές της και αυτό πιστεύω ότι είναι πολύ ε, σημαντικό. Είναι ένας τομέας στον οποίο πρέπει να γίνουν πολλές επενδύσεις. Εγώ θα ήθελα να κάνω κάποιο σχόλιο για τον τομέα των κατασκευών. Γιατί θα μπορούσαμε να έχουμε μεγάλη εξοικονόμηση στην ε, ε, κατασκευή ε, κυρίως κατοικιών. Χρειαζόμαστε περισσότερα κίνητρα και για τις νέες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτως ώστε ο τομέας ε, της οικοδομής ε, να αρχίσει να λειτουργεί καλύτερα ε, και με βάση νέα κίνητρα για ενεργειακή αποδοτικότητα. Δεν υπάρχουν πάντοτε τα κατάλληλα κίνητρα στον τομέα των οικοδομών και για την εξοικονόμηση θερμότητας ε, ε, και θα πρέπει να σκεφτούμε και τα οικονομικά κίνητρα τα οποία παρέχονται που διαφέρουν πάρα πολύ από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Θα μπορούσαν και τα διαρθρωτικά ταμεία να συνεισφέρουν δίνοντας οικονομικά κίνητρα προς τη σωστή κατεύθυνση. Άλλο ένα σημείο για το οποίο θεωρώ ότι η οδηγία είναι πάρα πολύ σημαντική στο πρώτο άρθρο, στην παράγραφο 3 και στο άρθρο 6 αναγράφονται ε, κάποια στοιχεία για τα οποία δεν είμαι απόλυτα βέβαιος ότι είναι στόχοι που μπορούν να τους επιτύχουν όλα τα κράτη-μέλη. Δεν είμαι βέβαιος ότι μπορούν όλα τα κράτη-μέλη να επιτύχουν αυτούς τους ετήσιους στόχους. Ευχαριστώ πολύ. Ε, κύριε Σένα. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ καλή ιδέα, ευγενής ιδέα θα έλεγα. Γιατί να δαπανούμε αφού μπορούμε να δράσουμε και να κάνουμε εξοικονόμηση στην ενέργεια. Για να εξοικονομήσουμε λοιπόν ενέργεια που είναι πολύ δαπανηρή και την οποία δεν την έχουν όλοι να σας πενθυμίσω. Άρα θα μπορέσουμε έτσι να καλύψουμε τις ανάγκες που δεν καλύπτονται αλλά και τις νέες, τις μελλοντικέ ανάγκες. Για μια ακόμη φορά όμως αυτή η ευγενής ιδέα εκτρέπεται και ωφελεί τελικά την κερδοφορία και ως το δυνατόν πιο σύντομα. Υπάρχει αγορά ενέργειας που θέλει να, κάνει, να βγάλει λεφτά. Θα υπάρξει ε, και το ίδιο πράγμα και στο μέλλον. Αν θέλουμε να κάνουμε οικονομίες θα πρέπει κατά προτεραιότητα να δούμε τους ε, τομείς που καταναλώνουν υπερβολική ενέργεια και να δούμε ποια παράστα είναι αυτά τα οποία ε, βγάζουν χρήματα με την ενέργεια και να ε, εφαρμόζονται οι κανόνες. Λοιπόν, ε, υπερβολική κατανάλωση. Με αυτά που προτείνουμε η κοινωνική στέγαση δεν επιδοτείται πλέον από τα ε, κράτη-μέλη και αυτοί οι οποίοι τελικά θα, θα πληρώσουν το βαρύτερο τίμημα για την εξοικονόμηση της ενέργειας θα είναι τα πλέον ευάλωτα νοικοκυριά. Θα πρέπει λοιπόν να επενδύσουμε στον τομέα αυτό για να έχουμε πραγματική εξοικονόμηση και οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν δυσκολίες να μπορέσουν και αυτοί να κάνουν τις οικονομίες. Το ίδιο και για τους ε, ιδιοκτήτες μικρών κατοικιών που δεν αξίζουν πάνω από 100.000 ευρώ. Δυσκολεύονται οι άνθρωποι αυτοί να πληρώσουν και τους φόρους τους κάτω από τα 1.000 ευρώ. Θα μπορούσαμε λοιπόν να έχουμε μία μείωση των φόρων κατά 25%. Αλλά δεν το κάνουμε, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Επομένως, οι εξοικονομήσεις θα γίνουν για κατηγορίες πληθυσμού που είναι ήδη πάνω από τα πρώτα. άρα δεν θα έχουμε και πολύ μεγάλη εξοικονόμηση. Θα πρέπει επίσης τα παράστα που κάνουν, βγάζουν χρήματα με τα χρήματα να τα καταπολεμήσουν. Πολύ περισσότερη ενέργεια αντιλάγει παρά παράχθηκε ε, πέρυσι, διότι πουλήθηκε η ίδια ενέργεια πολλές φορές και κάποιοι ενδιάμεση πλούτησαν από αυτό και εκεί πρέπει να κάνουμε εξοικονόμηση. Επίσης, να δράσουμε στην, ε, στο τομέα της παραγωγής. Όταν στο Κοινοβούλιο καθορίζουμε στόχους ώστε οι σιδηροδρομικές μεταφορές να είναι προτεραιότητα, τι διαπιστώνουμε. Διαπιστώνουμε ότι οι οδικές μεταφορές αυξάνονται σε βάρος των σιδηροδρομικών. Άρα εδώ έχουμε ένα πραγματικό πρόβλημα, πρόβλημα εξοικονόμησης ό,τι αφορά τώρα τη βιομηχανία. Πώς μπορούμε να καταλάβουμε ότι συνεχίζεται η μετεγκατάσταση παραγωγής σε χώρες που οι ίδιες έχουν ενεργειακό έλλειμμα στο όνομα της, του ανταγωνισμού ε, στο μισθολογικό. Τα 400 δις ευρώ που πηγαίνουν στην αγορά πρώτων υλών για την παραγωγή ενέργειας θα μπορούσαν αύριο μαζικά να ε, μειωθούν, αλλά χρηματοδοτικά η μάζα να αυξηθεί. Αν μια πρωτεΐλη είναι σπάνια, στην αγορά αυξάνεται και η τιμή της. Οπότε θα μπορούσαμε να έχουμε πάνω από 400 δις ε, ως δαπάνη, αφού θα είχαν αυξηθεί οι ε, κατώτατες τιμές. Επομένως, τι ερώτημα ε, τίθεται τι ζήτημα τίθεται. Αυτονομία, ενεργειακή αυτονομία στην ευρωπαϊκή επικράτεια. Όλες οι προποθέσει, όλοι οι όροι παραγωγής από αυτό το πρίσμα θα πρέπει να εξεταστούν. Ευχαριστώ. Κυρία Φαν Πολύ σύντομη θα είμαι, ούτε μισό λεπτό, Πρόεδρε. γιατί αυτό που είπατε κι εσείς έχει στρατηγική σημασία για όλους μας εδώ στο Κοινοβούλιο. Θέλουμε να έχουμε καλό αποτέλεσμα και δεν θα πρέπει να χάσουμε τη δική μας θέση υποτασσόμενη στη θέση του Συμβουλίου. Το Συμβούλιο έχει τη δική του θέση, εμείς έχουμε τις δικές μας θέσεις. Ας προσπαθήσουμε να ορίσουμε δεσμευτικούς στόχους και ας προσπαθήσουμε να έχουμε μια μεγάλη πλειοψηφία υπέρ των δικών μας θέσεων. Έχω εμπιστοσύνη προς τον εισηγητή και προς τους σκιώδεις εισηγητές και ιδίως προς τον σκιώδη εισηγητή της δικής μου ομάδας, συνάδελφος Μπένσον. Ευχαριστώ. Στην αρχή του 2011, 500 συνάδελφοι χαιρέτησαν την ψήφο τους ε, αυτή την πρωτοβουλία για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Τώρα, αν είμαστε διαιρεμένοι στην Ολομέλεια, τότε θα δώσουμε στην Κομισιόν ε, και στο ε, Συμβούλιο την ευκαιρία να επωφεληθούν και να εκμεταλλευτούν αυτή τη διαίρεση μεταξύ μας. Υπάρχει το θέμα της ισορροπίας. Υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να ε, παράγουν στην Ευρώπη. Ε, είδαμε και ότι ε, μέσω της ανακαίνησης μπορούμε να δημιουργήσουμε τοπικές θέσεις εργασίας και να υπάρχει κοινωνική συνοχή. Αλλά θέλω να επανέλθω σε αυτό που είπε ο κύριο Ζουρουμπή και τις μικρές και μεσές επιχειρήσεις. Έχουμε πολύ μεγάλη ανεργία αν ε, θέλουμε να αποφύγουμε την μεταγκατάσταση, αν ε, θέλουμε ε, οι άνθρωποι να μείνουν εδώ και να ζουν φυσιολογικά, θα πρέπει να δημιουργήσουμε και ένα νέο τεχνολογικό τομέα που θα εξάγει στις τρίτες αγορές. Εγώ νομίζω γιατί γι' αυτό το πρέπει να είμαστε ενωμένοι και όχι διαιρεμένοι όπως βλέπουμε σήμερα. Βουτιέρες παρακαλώ. Αν θέλετε. Ευχαριστώ. Εγώ έβαλα δύο είδη τροπολογιών. Θέλω να σας πω ότι είμαι απολύτως υπέρ της ε, μείωσης ε, της πατάλης ε, στα κτίρια αλλά εγώ θεωρώ ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί αυτή η οδηγία ως έχει. Δεν θέλω να είμαι αγγελοφόρος κακών μηνυμάτων, αλλά από ό,τι προβλέπω θα υπάρχει ε, πόλεμος μέχρι ε, τελικής πτώσης ε, στο Συμβούλιο. Είναι σημαντική στόχη, αλλά πού είναι τα μέσα για να φτάσουμε σε αυτούς τους στόχους. Όλοι θέλουμε να μειώσουμε, αλλά πού είναι τα μέσα, δηλαδή άρθρο 8. Πώς είναι δυνατόν ε, ε το χάρη ε, σε όλα τα σπίτια να έχουμε ένα νέο δίκτυο για να καταφέρουμε να πετύχουμε την ενεργειακή αποδοτικότητα. Πώς είναι δυνατόν σε πολλές πόλεις να έχουμε ένα εντελώ νέο σύστημα για να τις πηγές ενεργείας. Είναι αδύνατο με τις τεχνολογίες που έχουμε σήμερα και με τις προθεσμίες που έχουμε θέσει. Στην ΕΝΒΗ μόλις ψήφισα εκεί ε, περιόρισαν τις ε, προθεσμίες. Ε, δηλαδή, σε τρία χρόνια θα πρέπει να κάνουμε μία δύνατη επανάσταση. Χρειαζόμαστε στρατιές προσωπικού για να μετρήσουν την ενεργειακή αποδοτικότητα. Δεν έχουμε την τεχνολογία εγώ θα ήθελα να αλλάξω παραδείγματο χάρη το σύστημα θέρμανσης στο σπίτι μου, αλλά ε, δεν έχω τεχνολογία που να με το επιτρέπει. Και τι θα κάνω. Αυτό είναι το ένα. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να είμαστε πολύ σόφρονες με αυτή την οδηγία και θα έχουμε και τον κλασικό πόλεμο στο Συμβούλιο ε, γιατί δεν θέλουν να δαπανίσουν τα κράτη. Και επίσης, εγώ έχω και με πρωτοβουλία για το θέμα της ενεργειακής αποδοτικότητας στα ιστορικά κέντρα. Και έχουμε δύο λύσεις. Ε, ή θα δούμε το άρθρο 1, θα πάμε στο άρθρο 1, 3 μάλλον, τρία και ε, θα πρέπει να ζητήσουμε την αξιολόγηση της πολιτιστικής κληρονομιάς ή αυτό που νομίζω ότι θα είναι και πλέον σκόπιμο, θα είναι να υπάρχουν διαφορετικές λύσεις και διαφορετικοί δείκτες για τους ε, την πολιτιστική κληρονομιά και τα ιστορικά κέντρα. Πολλέ έρευνε γίνονται, αλλά δεν υπάρχουν αποτελέσματα. Αυτό που ζητάμε είναι να μην ε, βλάψουμε την πολιτιστική κληρονομιά και να έχουμε έτσι ξεχωριστούς δείκτες και ξεχωριστή αξιολόγηση, γιατί δεν μπορούν όλοι να φορέσουν το ίδιο κουστούμι. Μίλησαμε ε, για ε, ιστορικά κέντρα, ιστορικά σύνολα, έτσι εργαζόμαστε με τι πολιτιστικέ κληρονομιά. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο και στον κύριο Τούρμες και ζητώ και την κατανόηση της Επιτροπής γιατί περιμένουμε την Πολωνική Προεδρία που δεν μπορούμε να τους βάλουμε να περιμένουν. Πρέπει να δώσω το λόγο στον εισηγητή μετά από όλα αυτά. Κλοντ. Θα είμαι πολύ Θα είμαι πολύ σύντομος. Ε, νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε σήμερα το απόγευμα με τη συνάντηση των σκιωδών. Έτσι λοιπόν ε, δεν θα μπορέσω να απαντήσω σε όλους. Ε, κυρία Νέν, έχετε δίκιο ότι εδώ θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και την ανέχεια, την ενεργητική ανέχεια και έχουμε και τα άρθρα 5 και 6, έχουμε διάφορους μηχανισμούς εκεί, θα πρέπει να συναντηθούμε για να δούμε πώς ε, θα αντιμετωπίσουμε την ανέχεια και η Γαλλία έχει, έχει χρησιμοποιήσει τα διαφορετικά ταμεία για την ε, ανακαίνιση ε, στις εργατικές κατοικίες. Και μπορούμε να πάρουμε πολύ καλά παραδείγματα από τη Γαλλία. Και έτσι λοιπόν ε, φτάνω στο σχόλιο του κ. Μεζάρος. Νομίζω ότι έχετε δει και ο κυρίω στην Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη. Πρέπει να δούμε πώ ε, θα γίνουν επενδύσεις για να βελτιώσουμε τα κτίρια στις χώρες αυτές. Φυσικά αυτό έχει να κάνει με τη χρηματοδότηση και με τα διαρθρωτικά ταμεία, τα περιορικά ταμεία και την, και την κατάρτιση και γίνεται μια γέφυρα έτσι με αυτό που ο κύριος Ρούμπικ πρέπει να έχουμε επιτόπου μικρές μεσαίες επιχειρήσεις, μηχανικούς, αρχιτέκτονες που θα έχουν την κατάλληλη κατάρτιση. Και γι' αυτό στα άρθρα 13 και 14 προσπαθούμε να ενδυναμώσουμε και το στοιχείο της κατάρτισης. Και ο Πόλτη και ο Ιχιωτέν είπε ότι χρειαζόμαστε συνοδευτικά μέτρα και έχουμε το πρόγραμμα για την ΕΦΗ Ευρώπη στον τομέα τη ενέργεια. Εκεί κάνουμε ήδη αρκετά πράγματα για να προωθήσουμε την ενεργειακή αποδοτικότητα, την κατάρτιση κτλ. Και πρέπει να συνεχίσουμε. Γιατί τελικά δεν μπορεί κάποιος απλώς να νομοθετεί, χρειάζεται και ε, soft policies ε, για να συμπληρώσουν ε, τη νομοθεσία. Λοιπόν, μια ιδέα να αναφέρω οι ιδιωτικές τράπεζες στην Ευρώπη για τα επόμενα τρία χρόνια λάβουν ε, χρήματα χωρίς ε, ε, τέλος για 1% χωρίς να υπάρχει καμία προϋπόθεση, γιατί αυτό το αποφάσισε ο κ. Ντράγκη. Και επειδή βρισκόμαστε σε αυτή την παράλογη κρίση, ίσως αυτός είναι ο μόνος τρόπος να μπορέσουμε να πείσουμε τι ιδιωτικέ τράπεζε να αγοράσουν και πάλι κρατικά ομόλογα. όμω, γιατί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν ε, πρέπει να σέβεται τις ίδιους όρους με τις ιδιωτικές τράπεζες, γιατί δεν δίνουμε στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων επίσης 1% χρήματα χωρίς τέλος για να βοηθήσουμε να επενδύσει στην και αποδοτικότητα αλλά και σε υποδομές μεταφορών κτλ. Και νομίζω ότι αυτή η Επιτροπή πρέπει να συμβάλλει στην επίτευξη μια λύση. Γιατί αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι το εξή. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων λαμβάνει όλο ένα και μεγαλύτερο spread, ε, γιατί τελικά υπάρχει ποινικοποίηση από του οίκου αξιολόγηση ε, των μετοχών. Έτσι λοιπόν. Ε, αν έχουμε μείωση τη πιστοληπτική ικανότητα Γαλλία, τότε θα υπάρχει αύξηση ε, στα επιτόκια τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κυρία Καρβάλιο. Και νομίζω ότι απαντώ και στο θέμα της ε, συζήτησης για την, ε, τους στόχους ενεργειακής έντασης. Για όλες τις χώρες που έχουν ε, αρνητικές προβλέψεις για το ΕΕΠ, αν εισαγάγουμε ένα στόχο έντασης ενέργειας, οι χώρες αυτές θα βρεθούν σε μια αδύνατη κατάσταση, γιατί ακόμη και αν ε, το ήθελαν, δεν θα μπορούσαν να πετύχουν το στόχο. Και επομένω πρέπει να γεφυρώσουμε τη συζήτησή μας ε, και να δούμε και αυτά που είναι συνάδελφοι, Βίκη και άλλοι, να καταλήξουμε σε συμβασμό. Νομίζω και ο κύριος Γκέρεκ ε, αναφερθήκε σε αυτό το θέμα. Τώρα, οι ενεργοβόρες βιομηχανίες είναι κάτι διαφορετικό από τα κτίρια. Χρειαζόμαστε μία λύση και θα παρουσιάσω συμβιβασμό τον Ιανουάριο, όπου θα προσπαθήσω να βρω μια λύση χωρίς να δημιουργούμε φυσικά παραθυράκια, γιατί θέλουμε να φτάσουμε στο 20% και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ότι ο δείκτης ενεργικής έντασης ε, δεν ε, θα δημιουργήσει παραθυράκια κάποια κενά. Κύριε Κάλλη, κύριε Κέλλη, δεν ξέρω αν είστε ακόμα εδώ. Αλλά έχει δίκιο όταν λέει ο κ. Σκέλη ότι αυτές οι εταιρείε στην Ευρώπη που είναι επικεφαλής της αριστείας ε, στις ε, ε υπηρεσίες ε, θα βρουν αγορές στην Ασία, στη ΣΥΠΑ, στη Μέση Ανατολή κτλ. Μην πιστεύετε λοιπόν ότι εδώ μιλάμε μόνο για προϊόντα, αλλά μιλάμε και για υπηρεσίες, για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, για υπηρεσίες μηχανικής και θα μπορούσε να ε, ξαναδημιουργηθεί μια καλή αγορά υπηρεσιών στην Ευρώπη έτσι ώστε να κερδίσουμε εξαγωγικές αγορές. Μια ιδέα του Προεδρού που αναφέρει κύριε Φαμπρέντ, δεσμευτική στόχη έναντι δεσμευτικών μέτρων. Όταν ε, δείτε την έκθεσή μου και συγκεκριμένα την τροπολογία που κατέθεσα το Νοέμβριο, δημιούργησε ένα παράρτημα με λεπτομερείς εθνικούς ε, δεσμευτικούς στόχους. Και αυτό το έκανα μαζί με εμπειρογνώμονε και η Γερμανία θα πρέπει να είναι ικανοποιημένη γιατί ακριβώς αυτός κάνει και η Γερμανία στη χώρα της. Και το ίδιο κάνει μάλλον και το ίδιο υπέσχεται και η Γαλλία. Επομένω και αυτή πρέπει να είναι ικανοποιημένη. Αυτό το παράρτημα η Προεδρία της Δανίας μάλλον πήρε αυτό το παράρτημα, πήγε στο Βερολίνο και στο Λονδίνο και στο Παρίσι και στη Μαδρίτη. Και το αποτέλεσμα των πρώτων συζητήσεων της κυβέρνησης της Δανίας ήταν το εξή. Ότι όλες οι κυβερνήσεις είπαν «Α, εμείς σε καμία περίπτωση δεν θα πάμε προς αυτούς τους στόχους». Εγώ δεν έχω εγκαταλείψει αυτή την ιδέα, αλλά Όλοι εσείς ε, που θέλετε να είστε επαγγελματίες διαπραγματευτές, κοιτάξτε, θα προσπαθήσουμε να έχουμε όσο δυνατόν πιο δεσμευτικούς στόχους ως προς το 20%. Αλλά να ανοίξουμε τις διαπραγματεύσεις μόνο σε αυτό και είμαστε εντελώ ε, απογυμνωμένοι κατά τα λοιπά, αφήσουμε δηλαδή κατά μέρους όλα τα μέτρα, πώς θα διαπραγματευτούμε δεν θα έχουμε ε, θα είμαστε τελείω αποκοινωμένοι. Και εγώ όταν ήμουν ε, νέο, έπαιζα strip poker και πάντοτε φορούσα πάρα πολλά ρούχα. Ποτέ δεν πήγαινα γυμνό στο strip poker. Και ίσω ε, λοιπόν αυτό είναι ένα από του λόγου που προσπαθώ να είμαι καλό διαπραγματευτή. Κύριε Γκίρεκ, πρέπει να καθίσουμε από κοινού δεν ξέρω αν στην ακρόαση που είχαμε τους εμπειρογνώμονες. Στην ακρόαση κατέστησα φές ότι επειδή βρισκόμαστε σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, οι ευρωπαϊκές, ανατολικοευρωπαϊκές οικονομίες από σήμερα μέχρι το 2020 θα αναπτυχθούν 5-5,5-6% ε, ετησίως και πάλι όμως θα είναι κάτω από την βασική προβολή που έγινε το 2007. Νομίζω ότι έχουμε πρόβλημα. Πρέπει να εξηγήσουμε καλύτερα τι σημαίνουν στην πραγματικότητα τα στοιχεία της Κομισιόν. Νομίζω ότι λόγω της ύφεση είναι πιο εύκολο να πετύχουμε τους στόχους της Κομισιόν και εγώ θέλω ότι σεβαστώ. Τώρα είναι πιο εύκολο από το 2007. Αλλά έχω Όταν ε, μιλάω, βλέπετε πόση εμπειρία έχει στη διαπραγμάτευση. Έτσι λοιπόν, ε, ε, συμπαραγωγή. Έχετε δίκιο, δεν είναι το ίδιο με την τηλεθέρμανση και τη τηλεψήξη. Πρέπει να λάβουμε υπόψη και τη βιομηχανική συμπαραγωγή. Θα δούμε και αυτό το θέμα φυσικά, το πώς θα συμπεριλάβουμε τις ενεργοφόρες βιομηχανίες Δεν θα μπω στις λεπτομέρειες που αναφέρατε. Κυρία Χόλ. Για τις ε, δημόσιες συμβάσεις. Είναι δύσκολο θέμα. Γιατί, Γιατί αύριο, Τετάρτη, ο Επιτροπός θα παρουσιάσει ένα θεωρημένη οδηγία πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις. Ποια είναι η κατάσταση σήμερα. Όταν έχουμε δημόσια προσκλήση υποβολής προτάσεων, ε, επιτρέπεται μόνο να αγοράσει το φθηνότερο την ίδια τη στιγμή που αγοράζει. Και φυσικά αυτό είναι τεράστιο εμπόδιο. Αν αγοράσει ένα ψυγείο, δεν μπορεί να αγοράσει ένα ψυγείο τριπλό Α. Αλλά αν το ψυγείο αυτό είναι 5% πιο ακριβό από ένα άλλο ψυγείο που θα σου κοστίσει τελικά πολύ περισσότερα χρήματα κατά τη διάρκεια του κύκλου της ζωής του. Έτσι λοιπόν ε, αύριο ε, αυτή η προσέγγιση κύκλου ζωή υπάρχει σε αυτό το πλαίσιο που θα προσυστεί και θα πρέπει να συζητήσουμε και εμεί κάτι τέτοιο στο πλαίσιο τη οδηγία μα. Δηλαδή, αν ε, πέφτει το κόστο κύκλου ζωή, τι σημαίνει αυτό για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Θα σταματήσω εδώ, γιατί δεν έχουμε και χρόνο. Είναι πολύ σκληρή δουλειά, αλλά νομίζω θα τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λυπάμαι που δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά με συγχωρείτε. Είχατε, κύριε Τούρμε, ούτω ή άλλω μια μισή ώρα για τη συζήτηση αυτή. και έχουμε ήδη καθυστερήσει ένα τέταρτο. Τώρα θα επιδεχτούμε τον πρόσωπο τη Πολωνική Προεδρία. Υπάρχουν και κάποιοι που αποχωρούν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 να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης. Ε, έχουμε εδώ την τιμή να επιδεχόμαστε τον ε, κύριο Καλίνσκι, ο οποίος είναι υπεύθυνο ε, ενέργειας, εκπροσωπεί την Πολωνική Προεδρία, το γνωρίζουμε ήδη, δεν θα μακρηγορήσω εγώ. Θα σας παρακαλούσα να κάνετε λίγο ησυχία και όσοι αποχωρούν παρακαλώ χωρίς θόρυβο για να δώσουμε το λόγο στον κύριο Καλίνσκι για να μπορέσει να τοποθετηθεί. Καλώς ήρθατε κύριε Καλίνσκι, έχετε το λόγο. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή το ότι βρίσκομαι εδώ σήμερα για να σας παρουσιάσω εν συντομία ε, το έργο του Συμβουλίου στον τομέα της ενέργειας. Ε, μιλάω για το Συμβούλιο Μεταφορών Τηλεπικοινωνίων και Ενέργειας. Θα σας μιλήσω επίσης και για το έργο του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας ε, στον τομέα της βιομηχανίας για το διάστημα της Πολωνικής Προεδρίας. Καταρχάς όμως θα ήθελα να πω ότι δεν θα ήταν να μιλήσω για το έργο του Συμβουλίου χωρίς να αναφέρω τις προσπάθειες που έχει καταβάλει η Ουγγρική Προεδρία σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό στο διάστημα που προηγήθηκε. Και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο Ενέργειας ε, κατέληξαν σε συμπεράσματα τα οποία θέτουν ε, τις κατευθύνσεις ε, έθεσαν μάλλον τι κατευθύνσει για το έργο τη Πολωνική Προεδρία στο τομέα τη ενέργεια από την περίοδο του Ιουλίου έως το Δεκέμβριο 2011 δύο ήταν τα θέματα που θέσαμε ως προτεραιότητα. Εξωτερική ενεργειακή πολιτική και οδηγία για την ενεργειακή απόδοση. Σε ό,τι αφορά το πρώτο ζήτημα, που ήταν ε, και βασικό κομμάτι της, ε, του προγράμματος της Πολωνικής Προεδρίας. Ε, στις 24 Νοεμβρίου το Συμβούλιο με τα συμπεράσματά του ενισχύει την εξωτερική ενεργειακή πολιτική. Οι διαπραγματεύσεις ήταν δύσκολες ό,τι αφορά το περιεχόμενο των συμπερασμάτων. Και αυτό δείχνει πόσο αναγκαία είναι για την Ευρωπαϊκή Ένωση μια συνεκτική και αναρμονισμένη προσέγγιση. Δείχνει πόσο επίγον είναι να ενισχυθεί η δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μιλά στο διεθνές προσκήνιο με μια φωνή. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στα βασικά στοιχεία των συμπερασμάτων του Συμβουλίου Μεταφορών Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας, που ενέκρινε και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 9 Δεκεμβρίου. Πρώτα απ' όλα, ενίσχυση του συντονισμού στην εξωτερική ενεργειακή πολιτική. Πρέπει να βρούμε τα μέσα, τα εργαλεία, τις δομές που θα βοηθήσουν να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, διατηρώντας και τη διάκριση αρμοδιοτήτων μεταξύ θεσμικών οργάνων της Ένωσης και κρατών μελών και μεταξύ θεσμικών οργάνων βάσει των συνθήκων. Επίσης, πρέπει να ενισχύσουμε το σύστημα συντονισμού, ιδίως σε ό,τι αφορά την ε, καθιέρωση κοινών θέσεων μεταξύ κρατών μελών και Συμβουλίου. Αυτό θα πρέπει να πραγματοποιείται με τακτικές συναντήσεις ε, του Αρμόδιου Συμβουλίου και οι συναντήσεις των ε, γενικών ε, διευθυντών που θα συζητούν τις στρατηγικές πτυχές και τις πολιτικές πτυχές. Επίσης, δημιουργία ενός καταλόγου διεθνών οργανισμών με τους οποίους θα έχουμε συντονισμό. Επίσης, ενίσχυση της ενεργειακής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ σημαντική πτυχή γιατί θα μας επιτρέψει να έχουμε ανταγωνισμό, βιώσιμη ανάπτυξη και ασφαλή ενεργειακό εφοδιασμό. Αυτά είναι τα τρία βασικά σημεία. Σε πνεύμα αλληλεγγύης θα στηρίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης οποιοδήποτε κράτος μέλος με την παρουσία της Επιτροπής στις διαπραγματεύσεις, αν αυτό ζητηθεί, στις διαπραγματεύσεις, διμερείς διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες. Επόμενο. Πρέπει να δοθεί νέα όθηση στην επέκταση της ενεργικής κοινότητας και την ε, συνθήκη του για τον ενεργειακό χάρη. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών με βάση την εσωτερική ενεργειακή αγορά με τη μορφή της συνεργασίας και της εναρμόνισης των κανονισμών και των ρυθμίσεων που διέπουν τις σχέσεις με τις γειτονικέ χώρες. Επίσης, ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας με την ανάπτυξη των σχετικών υποδομών. Μεγαλύτερη ασφάλεια επίσης ε, στη, στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας, αλλά και στις εξέδρες ε, εξόριξης. Ένα άλλο θέμα είναι οι αρχές που θα πρέπει να διέπουν τι συμφωνίες εταιρική σχέση που συνάπτουμε με τρίτες χώρες και επίσης θα πρέπει να συμφωνήσουμε για την ανάληψη νέων πρωτοβουλειών για στρατηγική σχέση με ΙΠΑ, Ινδία, Ρωσία, Κίνα, Νότια Αμερική και Βραζιλία. Ιδίω, με τη Ρωσία η νέα συμφωνία είναι ένα θέμα στο οποίο εστιάζουμε, όπως και ο δικός χάρτης για τη συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας μέχρι το 2050. Μία από τις βασικές αποφάσεις είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφώνησε να εγγυηθεί τη στήριξη των κρατών μελών στις διμερείς διαπραγματεύσεις που θα έχουν για ενεργειακά θέματα. Ήδη στο Συμβούλιο έχει ξεκινήσει η σχετική εργασία συγκεκριμένα ανταλλαγή πληροφοριών, σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών για τις διακυβερνητικές διαπραγματεύσεις. Αυτό θα διευκολύνει την επίτευξη συμφωνίας με τους ε, μείζονες ε, προμηθευτές ενέργειας. Είμαι βέβαιος ότι σε στενή συνεργασία με το Κοινοβούλιο, με το οποίο ήδη συνεργαζόμαστε σε άλλες προτάσεις, σε άλλα σχέδια, επιδανικής προεδρίας θα έχουμε πλήρη επιτυχία σε αυτό το φάκελο. Μια άλλη προτεραιότητα της εξάμηνης αυτής περίοδου για την Προεδρία μας ήταν η επεξεργασία της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση. Η Πολωνική Προεδρία έχει κάνει εντατική δουλειά και τώρα μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ένα κείμενο που έχει προχωρήσει και αντικατοπτρίζει την κατάσταση στο Συμβούλιο. Όπως είδαμε και στην έκθεση προόδου του Συμβουλίου Τηλεπικοινωνιών ε, Τεχνολογιών ε, στις, ε, το Νοέμβριο συγκεκριμένα. Η Πολωνική Προεδρία λοιπόν έχει σημειώσει πρόοδο στο νομοθετικό αυτό κείμενο για να είναι πιο ευέλικτα τα μέσα και οι μηχανισμοί που προτείνει η Κομισιόν, ενώ ταυτόχρονα φροντίζει να διατηρηθεί η φιλοδοξία, ο βαθμός φιλοδοξίας για τη δημιουργία αυτού του ευέλικτου πλαισίου. Στόχος είναι να έχουμε 20% μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση μέχρι το 2020. Η Προεδρία θεωρεί ότι το παρόν κείμενο είναι μια καλή βάση εργασίας για την επόμενη Προεδρία, ώστε να έχουμε αρκετά νωρίς διακυβερνητική συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, κάτι το οποίο ζητά και στα συμπεράσματα της 9ης Δεκεμβρίου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το, η Πολωνική Προεδρία σημειώνει με ικανοποίηση την συνέχεια των εργασιών για την ολοκλήρωση των εσωτερικών αγορών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου μέχρι το 2014. Επίσης, τα κράτη-μέλη καταβάλουν προσπάθειες στον τομέα αυτό. Το ίδιο και η Εθνική Ρυθμιστική Φορείς και οι διαχειριστές δικτύων. Γίνονται προσπάθειες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους οργανισμούς Άσερ και Έντσο. Με όλα αυτά θα δημιουργηθεί τελικά μια εναρμονισμένη ε, αγορά, διατάξει την εναρμονισμένη αγορά. Θα προωθηθούν περιφερειακές πρωτοβουλίες, η περιφερειακή ολοκλήρωση των αγορών, ενώ θα εισαχθεί και νομοθεσία για την ενιαία εσωτερική αγορά χάρη στις ε, πολύ σημαντικές προσπάθειες της Ουγγρικής Προεδρίας, καταφέραμε και εμείς από πλευράς μας να ολοκληρώσουμε γέρο τις δικές μας εργασίες με το πρόγραμμα REMIT. Έχουμε επίση ε, συνεχεί σταθερέ διαβουλεύσεις με τα κράτη-μέλη, ιδίω για περιπτώσει όπου οι αποφάσει οι θα μπορούσαν να επηρεάσουν το ενεργειακό μείγμα ή τι ενεργειακέ ε, δυνατότητε ε, τη μιας ή της χάλης χώρας. Οι υποδείξεις, προτάσεις που διατυπώνονται στις συνεδριάσεις που οργανώνει η τη αλλη χωρα οι υποδειξεις προτάσει που διατυπωνονται στις συνεδριάσει χάρη πολωνικη προεδρια παραδειγματο συνάντηση των Υπουργών ενέργεια το Σεπτέμβριο στο Βρότσλαφ, δείχνουν και έχουν δείξει και στο παρελθόν ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει το σχετικό ζήτημα πολύ άμεσα. Θα ήθελα επίσης κύριε και κύριοι να επιστήσω την προσοχή σας σε κάποιες άλλες προτάσεις που έχουμε συζητήσει στο Συμβούλιο. Πρώτα απ' όλα, σχέδιο κανονισμού για τα κατευθυντήριες γραμμές για τι Ευρωπαϊκέ Ενεργειακέ υποδομές. Οι Υπουργοί Ενέργεια συνεδρίασαν δύο φορές, ανεπίσημη συνάντηση 19 Σεπτεμβρίου και ανεπίσημο συμβούλιο 24 Νοεμβρίου. Και εκεί συζήτησαν το μέλλον των διευρωπαϊκών δικτύων στον τομέα τη ενέργειας. Αμέσως μετά την πρόταση της Κομισιόν άρχισε εντατική εργασία το Συμβούλιο στην ομάδα εργασίας της σχετική για αυτό το θέμα. Επόμενο, Επόμενο σχέδιο. Δημοσίευσε το Συμβούλιο σχέδιο κανονισμού για την ασφάλεια των ε, εξεδρών ε, εξόρισης, γεώτρησης. Ε, είδαμε την καταστροφή που είχαμε στο κόλπο του Μεξικού το 2010 και θέλουμε να αποτρέψουμε τέτοιες καταστροφές στο μέλλον. Τώρα, τους επόμενους μήνες πρέπει να σας πω ότι θα έχουμε πολύ εντατική δουλειά και ε, εμείς στο Συμβούλιο αλλά και το Κοινοβούλιο. Πολύ σημαντικοί μήνες λοιπόν, αν θέλουμε να ενισχύσουμε την ενιαία στερική αγορά, αν θέλουμε να αγγιηθούμε την βιώσιμη, την αηφόρα ανάπτυξη, αλλά και την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Δράτω με τις ευκαιρίες για να ευχηθώ στους δανούς συναδέλφους μου από το Συμβούλιο κάθε επιτυχία στη δουλειά τους όσο θα προεδρεύουν των συνεδριάσεων του Συμβουλίου. Γνωρίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στον κύριο Παύλακ, τον Υπουργό μου και σε μένα προσωπικά έχει παράσχει κάθε υποστήριξη. Και ελπίζω και εμείς να έχουμε επιτελέσει το έργο μας ε, σωστά και να είχαμε ποδοτική διοργανική συνεργασία. Εν συντομία τώρα να σας μιλήσω για το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και συγκεκριμένα το σκέλος της βιομηχανίας. Δύο εμβληματικές πρωτοβουλίες ε, προωθήσαμε στο πλαίσιο της στρατηγικής στην Ευρώπη του 2020. Πρώτα απ' όλα την ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική στον τομέα, ε, στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και πώς μπορούμε ε, να αξιοποιούμε τους πόρους μας. σε ανακοινώσεις που εκδόθηκαν φέτος. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σας πω πόσο σημαντική είναι η βιομηχανία για την ευημερία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τη θέση της Ευρώπης να είναι ένας πρωταγωνιστής σε παγκόσμιο επίπεδο και πηγή καινοτομίας. Από τότε που πρωτοδημοσιεύτηκαν τα σχετικά έγγραφα ένα χρόνο πριν, έχουμε περάσει τώρα στη φάση της υλοποίηση των προτάσεων αυτών στην Ευρώπη. Αν δείτε τη δέσμη μέτρων για την τυποποίηση, βλέπετε κάποια δείγματα της πρόοδου που έχουμε σημειώσει, όπως και την ανακοίνωση που είχαμε για το Small Business Act, που στόχο έχει την διεθνοποίηση των ΜΜΕ και τη μεγαλύτερη εταιρική ευθύνη. Προσπαθήσαμε να υπογραμμίσουμε την ε, σημασία της βιομηχανίας δεδομένων και των σημαντικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε. Επομένω, στις 29 Σεπτεμβρίου τα συμπεράσματα για την ανταγωνιστική ευρωπαϊκή οικονομία τονίζουν την ε, αποφασιστικότητά μας ε, να εγγυηθούμε μια συνέχεια κανονιστική και μια προβλεψιμότητα για τις επιχειρήσεις. Το Συμβούλιο υπογράμμισε την Συμφωνία της Ανταγωνιστικότητας και της Μελέτης Επιπτώσεων των νέων νομοθετικών προτάσεων στον ε, τομέα αυτό. Πρέπει λοιπόν να αξιοποιήσουμε τα μάλα του σπόρους και τις πηγές, τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για να εξασφαλίσουμε την ευημερία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως είπα, το Συμβούλιο τόνισε τη σημασία που έχει η αξιολόγηση των επιπτώσεων της νομοθεσίας ε, για την ανταγωνιστικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί και ο άμεσος αντίκτυπος είναι σημαντικός και ο έμεσος αντίκτυπος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διατυπώσει μια πρόταση για την απόδειξη το competitiveness proofing. Στις, ε, την 21 Νοεμβρίου συναντήθηκε η υψηλή ομάδα, υπομάδα υψηλού επίπεδου για την ανταγωνιστικότητα για να δώσει πνοή σε αυτή την πρωτοβουλία. Και είπαμε ότι ένα τέτοιο κείμενο θα πρέπει να εφαρμοστεί και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στις αρχές Δεκεμβρίου το Συμβούλιο υιοθέτησε τα συμπεράσματά του για την υιοθέτηση της εμβληματικής ε, πρωτοβουλίας για τη βιομηχανία. Έχουν ήδη αναλυφθεί κάποιες δραστηριότητες στον τομέα αυτό και στον τομέα της εταιρική ευθύνη και της διεθνοποίησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τελέσαμε νομίζω περαιτέρω πρόοδο στα θέματα αυτά. Σε ό,τι αφορά την προστασία των δημιουργών βιστεχνία, την καταπολέμηση τη γραφειοκρατία και την βελτίωση τη ανταγωνιστικότητα. Ένα χρόνο μετά βέβαια έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις ίδιες προκλήσεις στην Ευρώπη. Και μπορείτε να δείτε ότι δεν υπάρχει ε, μεγάλη εμπιστοσύνη στην οικονομία και ίσως επιδεινωθούν ακόμη περισσότερο οι προοπτικές η κατάσταση των χρηματοπιστωτικών αγορών δεν είναι καλή, χρειάζεται δημοσιονομική εξυγίανση και σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να προωθηθεί ταυτόχρονα και η οικονομική ανάπτυξη. Δεν θα πρέπει όμως ταυτόχρονα να επιτρέψουμε τη λήψη αποφάσεων που θα παρακολύσουν την οικονομική ανάκαμψη. Θα πρέπει να δεχθούμε το γεγονός ότι ίσως το επόμενο έτος να μην έχουμε και κάποια σημαντική βελτίωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της θα πρέπει ίσως να λάβουν και περαιτέρω δράση για να εγγυηθούν την ανταγωνιστικότητα στη βιομηχανία, για να βελτιώσουν την οικονομική ανάπτυξη και επομένως έτσι να συμβάλλουν και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Η Προεδρία αυτή νομίζω ότι έχει δώσει και κάποιες ελπίδες ότι είναι εφικτή η στόχη αυτή. Επιτελέσαμε θετικό έργο και αυτό χάρη στο κλίμα, στην ατμόσφαιρα που επικράτησε στις συζητήσεις. Τον Ιούλιο είχαμε συζητήσεις με τη βιομηχανία στο Σόποτ και στο Γκτάνσκ το Σεπτέμβριο είχαμε μια συνεδρίαση για την κοινωνική εταιρική ευθύνη. Τον Οκτώβριο στην Κρακοβία συναντηθήκαμε με μικρομεσαίες επιχειρήσεις και συζητήσαμε ε, τον τρόπο εμβάθυνσης της ενιαίας αγοράς. Ελπίζω να συνεχιστεί η συνεργασία αυτή. Κοινή είναι η στόχη. Η Ευρώπη χρειάζεται ισχυρή ε, καινοτόμα βιομηχανική βάση Ολοκληρώντα, κύριε και κύριοι, θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Επιτροπής ΙΤΡΕ, τον κύριο Χέρμπερτ Ρόιλ, για την υποστήριξη που παρήχε στο έργο μας. Θα ήθελα επίση να ευχαριστήσω τους αντιπροέδρους αλλά και όλα τα μέλη της Επιτροπής ΙΤΡΕ. Χωρίς τη δική σας δέσμευση, αφοσίωση και συνεργασία, δεν θα είχαμε επιτύχει το έργο μας ως Πολωνική Προεδρία. Ευχαριστώ. Ανταποδίδω και εγώ τις ευχαριστίες ε, κύριε Καλίσκη. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που συνεργάστηκαν με την ε, Πολωνική Προεδρία και πρέπει να σας πω ότι ε, όλοι οι συνάδελφοι που συνεργάστηκαν με την Πολωνική Προεδρία ξέφρασαν ότι ήταν ιδιαίτερα υποστηρικτικοί και πάντοτε τονίζει η Πολωνική Προεδρία ότι η βιομηχανία στην Ευρώπη έχει ένα κοινό μέλλον. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το λαμβάνουν υπόψη οι πολιτικοί θύνοντες ε, όταν λαμβάνουν οι πολιτικοί τις αποφάσεις. Και πριν έρθετε ακριβώς είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Βλέπω ότι ήδη υπάρχουν κάποιοι ομιλητέ, Κυρία Χίμπνερ. Ευχαριστώ πολύ. Ο Υπουργός τόνισε πολλές φορές το ρόλο της Προεδρίας για την βιομηχανική πολιτική, για την πολιτική για το ενεργειακό μείγμα και για την ε, πολιτική για την ε, ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Στη διάσκεψη κορυφής ε, στο Ντέρμπαν συζητήθηκαν, συζητήθηκαν θέματα με σημαντικές επιπτώσεις και στην οικονομική μας ανάπτυξη. Η ερώτησή μου είναι τι επιπτώσεις θα έχουν οι δεσμεύσεις του Ντέρμπαν για την ευρωπαϊκή οικονομία, εφόσον μιλάμε και για μείωση εκπομπών. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσω το λόγο στον κύριο Καλίσκη ή να δώσουμε το λόγο στον κύριο Γκίρεκ που είχε ζητήσει το λόγο. Ας ακούσουμε και τον κύριο Γκίρεκ πρώτα. Ευχαριστώ. Έχω δύο ερωτήσεις. Η μία αφορά το ενιαίο σύστημα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Πολλοί επενούν την Πολωνία και ο κύριος Μπαρόζο επένεσε την Πολωνία ε, για την ε, επιτυχία την οποία είχε στους τομείς αυτούς που συζητάμε. γίνονται και κάποιες τροποποίησεις στον κανονισμό και συζητείται το 50% συμμετοχής για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Πώς θα προσδιοριστεί η αγορά, θα ορίζεται η αγορά βάσει του αριθμού κατοίκων ή με βάση κάποιο διαφορετικό δίκτυο. Και έχω και άλλη μια ερώτηση. Μια ερώτηση που έκανα και προς τον εισηγητή για τα θέματα ενεργειακής απόδοσης και δεν έλαβα απάντηση. Θέλω να ρωτήσω εάν είναι δυνατόν μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αυξήσει κατά το 20-30% την ενεργειακή της απόδοση, αλλά παράλληλα να αυξάνει και την κατανάλωση ενέργειας αντίστοιχα. Είναι κάτι το οποίο είναι πιθανόν. Κύριε Καλίσια, έχετε το λόγο για να απαντήσετε. Ας ξεκινήσω με τις κυρίες, ε, την ερώτηση που μου έκανε η κυρία Χίμπνερ. Αν δείτε τις οικονομίες των κρατών μελών μεμονωμένα, ή την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, οι μονομερείς δεσμεύσεις μειώσεων δεν θα ωφελήσουν την ε, οικονομία μας αν δεν κάνουν το ίδιο και οι άλλες χώρες. Διαφορετικά θα μειώσουμε σημαντικά την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας ε, λόγω του φαινομένου που αποκαλούμε carbon leakage, ε, τη μετεγκατάσταση δηλαδή βιομηχανιών από την Ευρώπη προς άλλες χώρες λόγω των μειώσεων που κάνουμε εμείς στις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος. Στο Durban συμφώνησαν όλες οι χώρες ότι μέχρι το 2015 θα καταλήξουν σε μία συνολική συμφωνία που θα καλύπτει όλες τις χώρες του πλανήτη και τις αναπτυσσόμενες χώρες και θα επιβληθούν στόχοι μείωσης σε όλες τις χώρες ανάλογα με τα επίπεδα εκπομπών κάθε χώρας. Ο συντονισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε πολιτικό και σε τεχνικό επίπεδο ε, Μα έδωσε τη δυνατότητα να εκφραστούμε με μία και μόνη φωνή στον Τέρμπαν και αυτή η ενότητα απόψεων ε, ήταν προ όφελο της Ευρωπαϊκή Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατόρθωσε να εκπληρώσει το στόχο της βάσει της εντολής που δόθηκε από το Συμβούλιο Περιβάλλοντος του Οκτωβρίου. Και αυτή η απόφαση δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μελλοντικές συμφωνίες και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει οι χώρες που καλύπτονται από τη συμφωνία να επιτύχουν τους στόχους τους. Η επιτυχία λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγκυται στην ισορροπημένη προσέγγιση για την μελλοντική συμφωνία για τη συνέχιση του πρωτοκόλλου του Κιώτο. Και τώρα προς τον κύριο Γκίρεκ. θα μπορούσε κανείς να απαντήσει το εξής στην ερώτησή σας για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Η απάντηση είναι ναι, μπορούμε να αυξήσουμε την ενεργειακή αποδοτικότητα, ενώ παράλληλα μπορούμε και να αυξάνουμε την κατανάλωση ενέργειας. Η Πολωνική Προεδρία προσπάθησε να συνεχίσει τις εργασίες σχετικά με τη δέσμη μέτρων για την ενεργειακή αποδοτικότητα, τηρώντας και τις συμβιβαστικές λύσεις τις οποίες έχουμε καταλήξει μετά από πολλά χρόνια διαπραγματεύσεων. έγινε πιο δύσκολο το έργο μας γιατί δεν ε, ήταν παρούσες η Ιταλία και η Ισπανία αλλά πιστεύω ότι τελικά η λύση την οποία επιτύχαμε είναι μια λύση που μπορεί να γίνει αποδεκτή. Και χάρη σε αυτή τη λύση στην οποία καταλήξαμε, η Ιταλία έχει εκδηλώσει την προθυμία της ε, να συμμετάσχει σε αυτή την πρωτοβουλία και για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και γιατί θα αποτελέσει απλούστευση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η συμβαστική λύση μιλά για διπλώματα ευαισθητεχνία σε τρει γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά και ήταν ένα από τα πιο ευαίσθητα θέματα που χειριστήκαμε κατά την Προεδρία μας. Αυτό το σύστημα που βασίζεται στις τρεις γλώσσες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας ήταν η μόνη λύση στην οποία μπορούσαμε να καταλήξουμε μια λύση που να είναι αποδεκτή από όλους. εάν δεν υπάρξει συμφωνία θα πρέπει να ακολουθήσουμε τη διαδικασία συντονισμού. Θέλω να πω ότι η συνεργασία μεταξύ των οργανισμών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας θα είναι μια καλή λύση για τις χώρες που δεν έχουν μεγάλη δραστηριότητα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Συνολικά πιστεύω ήταν μια θετική λύση. Ο κύριος э, Ευχαριστώ. Έχω μια πολύ σύντομη ερώτηση. Έχουμε πολλές εκθέσεις εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχέση με το κλείσιμο των αρχείων. Ξέρω πόσο σημαντικό είναι ο άνθρακάς στην Πολωνία, ο Λιγνίτης. Έτσι λοιπόν θέλω να ρωτήσω σχετικά με τα αποτελέσματα της Πολωνικής Προεδρίας για τις τεχνολογίες που δεν θα παράγουν τόσο υψηλές εκπομπές άνθρακα. Odpowiadając na to pytanie, potwierdzę e, stwierdzenie. Να επιβεβαιώσω καταρχήν τα όσα είπατε για την σημασία του Λιγνίτη για την πολωνική οικονομία, αλλά και όχι μόνο για την πολωνική οικονομία. Ένα πρόβλημα που έχουμε είναι ο ορισμός ε, του καθαρού άνθρακα. Δηλαδή, θέλουμε να αυξήσουμε την ε, παραγωγή ενέργειας από 23% ή από 45% σε 60%. Με, λύσαμε. Ε, για το μελλοντικό δικό χάρτη για την ενέργεια μέχρι το 2050. Αυτό συζητείται τώρα στην ομάδα υψηλού επίπεδου. Και πιστεύουμε ότι η προώθηση των ε, τεχνολογιών με χαμηλές ε, εκπομπές άνθρακα, ανεξάρτητα από το πώς θα τις ορίσουμε, είναι ένα ουσιαστικό τμήμα της ενεργειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, συζητήσαμε σε πολλά βήματα αυτό το θέμα κατά καθ' όλη τη διάρκεια της Πολωνικής Προεδρίας. Δεν υπάρχουν άλλοι ομιλητέ. Κλείνουμε λοιπόν αυτό το σημείο τη σημερινή διάταξη. Θέλω να ευχαριστήσω τον καθηγητή Καλίσκη. Σα ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και την πολωνική κυβέρνηση Προσωπικά θεωρώ ότι ήταν εξαιρετική η περίοδος της Πολωνικής Προεδρίας. Είχαμε πολύ καλή συνεργασία. Κατορθώσαμε να καταλήξουμε σε αποτελέσματα, σε πολλά και σημαντικά θέματα. Και συνεισφέρατε ε, στην ευρωπαϊκή πολιτική συζήτηση ώστε να υπάρχει ε, και ρεαλισμός και να ληφθούν υπόψη τα συμφέροντα της βιομηχανίας. Πολύ χρήσιμη η συμβολή σας και ελπίζω ότι οι καρποί των εργασιών σας θα μας συνοδεύουν και στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν και για την παρέμβασή σας και παρακαλώ να μεταβιβάσετε τις ευχαριστίες μας και στους συνεργάτες σας. Ευχαριστώ πολύ. Και πάλι θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο για τη συνεργασία του. Και επίση θέλω να ευχαριστήσω και τα μέλη τη Επιτροπή για τη βοήθειά του. Γιατί χωρί τη δική σα υποστήριξη δεν θα είχαμε μπορέσει να πετύχουμε τι προτεραιότητέ μα και του στόχου μα. Έτσι λοιπόν, από τα βάθη τη καρδιά μου και εκ μέρου της Προεδρίας, θέλω να ευχηθώ στην επόμενη Προεδρία της Δανίας καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ. Ε, πέρα στη συνεδρίαση λοιπόν και έχουμε πει ότι θα συναντηθούμε για ένα ποτήρι μιας και τελειώνει η χρονιά και έχουμε την ε, ευγενή πρόσκληση προς όλους. Ευχαριστώ πολύ.